Ακούτε την ελληνική καμπίνα παρακαλώ. Εντάξει, λειτουργεί τώρα το σύστημα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Σας προτείνω στο σημείο 11 της ημερησίας διάταξης να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ερικ Αλμπέρ, ιδρύτη του Γαλλικού Ιδρύματος ε, σχετικά με το στρες στην εργασία, στην ατομική και τη συλλογική του διάσταση. Πρόκειται για τις απόψεις που λάβαμε υπόψη κατά την εξέταση της σχετικής έκθεσης στο πλαίσιο της στρατηγικη 2007 2007-2012 για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Κύριε Έλμπερ, έχετε το λόγο για την παρουσίαση σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να περάσω στο, στην επόμενη διαφάνεια. Θα προσπαθήσω να σας δείξω ότι πέρα από το ίδιο το στρες, το μέγιστο ζήτημα που τη σήμερα μου φαίνεται στις επιχειρήσεις είναι ένα ζήτημα εργασιακών σχέσεων. Το στρες ε, είναι απλά μια πρόφαση για να μιλήσουμε για τις εργασιακές σχέσεις. Για να ξεκινήσουμε θα ήθελα ενώπιον αυτού του αξιοσέβαστου οργάνου ε, να επιστήσω την προσοχή σας ε, ότι το στρες αποτελεί ένα ιδεολογικό θέμα από την ουσία του. Ε, γιατί, διότι σε αυτό συναντώνται μια σειρά από, περιορισμοί, με συγχωρείτε που τόσο, καθυστέρησα τόσο πολύ, αποτέλεσε έναν παράγοντα στρες για μένα, υπήρχε πολλοί κόσμος κάτω, ε, κυκλοφοριακή συμφόρηση, πολλοί περιορισμοί που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το στρες, το οποίο αποτελεί ατομική υπόθεση, είναι το άτομο ενώπιον του περιορισμού, της πίεσης. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν με την πίεση πρέπει να μειώσουμε, να ελαττώσουμε τις ποιώσεις και να ρωτιέμαι τι κάνει η πόλη των Βρυξελών για να υπάρχουν λιγότερε κυκλοφοριακές συμφορήσεις το πρωί όταν κάποιος προσπαθεί να έρθει στη δουλειά του στο κοινοβούλιο, πώς γίνεται να έχουμε λιγότερες ουρές για να μπούμε στο κτίριο. Αυτή είναι λοιπόν η συλλογική άποψη του στρες, πρέπει να μειώσουμε τις πιέσεις Ορισμένα άτομα προσαρμόζονται καλά, άλλοι λιγότερο καλά και πρόκειται για μια ατομική υπόθεση. Λοιπόν, όταν κανείς προσαρμόζεται καλά, το πρόβλημα επιλύεται και ο άνθρωπος απελευθερώνεται από το στρες. Το στρες ε, περιλαμβάνει και μια ιδεολογική πτυχή. Αυτός είναι ένας ε, λόγος ε, για τον οποίο δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά αυτό το θέμα. Θεωρείται ότι όλοι μιλούσαν από άποψη πίεσης ή από ατομική άποψη. Ε, έτσι βλέπετε τις διάφορες αντιπαραθέσεις ε, ε, μεταξύ των θέσεων της πίεσης και της ελευθερίας του ατόμου. Με αυτό το σχεδιάγραμμα προσπαθώ να σας δείξω αυτό που μου φαίνεται πολύ σημαντικό για το στρες, οι πολλαπλές διαστάσεις του στρες. Στην επάνω γραμμή έχετε τρεις στήλε. Βλέπετε, έχουμε τους παράγοντες προβλέψεις μετά έχουμε τις συναλλαγές και μετά τα αποτελέσματα, τις συνέπειες οι παράγοντες πρόβλεψη είναι οι παράμετροι με τι οποίε μπορούμε να προβλέψουμε τι συνέπει στην κατάσταση στρε σε ένα άτομο. Αυτοί οι παράγοντε πρόβλεψη περιλαμβάνουν όπως βλέπετε πέντε ε, πλαίσια. Το πρώτο αφορά τα κοινωνικά, δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα. Εάν είστε μια γυναίκα με χαμηλό εισόδημα ε, μόνη της με παιδιά, ο παράγοντας πρόβλεψης είναι πολύ ανώτερος ε, από έναν άντρα παντρεμένο και με υψηλά εισοδήματα. Επίσης υπάρχουν οι πτυχές προσωπικότητας και γενετικές. Όλοι έχουμε μία ε, γενετική κληρονομιά η οποία μας προδιαθέτει και χαρακτηριστικά προσωπικότητας που μας προδιαθέτουν ε, στο να έχουμε λιγότερο ή περισσότερο στρες. Τέλος, ε, έχουμε τα, αυτά που ονομάζουμε life events, τα γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου, διάφορα γεγονότα, διάφορα συμβάντα, ένα παιδί άρρωστο ή προβλήματα στο ζευγάρι ή μόλις ε, πάθαμε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και αυτά μπορούν να μας προκαλέσουν περισσότερο ή λιγότερο στρες. Ε, τα χαρακτηριστικά σε αυτά τα τρία πλαίσια είναι ότι δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, τα υφιστάμεθα. Υπάρχει ένα κομμάτι του στρες το οποίο υφιστάμεθα και το οποίο δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καθόλου. Τέλ, στη συνέχεια έχουμε το επαγγελματικό στρες πώς βλέπετε στο τρίτο πλαίσιο. Αυτό μας ενδιαφέρει και μετά ένα πλαίσιο το οποίο αφορά τις συνθήκες ζωής, αν κάποιος αθλείται, αν έχει φίλους, ε, αν κοιμάται καλά το βράδυ, αν τρέφεται καλά. Ε, διάφορα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε και πολλές φορές δεν τηρούμε. Ε, αυτές οι δύο διαστάσεις λοιπόν, οι συνθήκες ζωής και η επαγγελματική ζωή είναι τομείς στους οποίους μπορούμε να δράσουμε συλλογικά και ατομικά. Στην τρίτη στήλη βλέπετε τις ε, συναλλαγές, τα transactions, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το στρες, αυτό που είναι καθοριστικό σε αυτό το τομέα, είναι ο τρόπος ταυτόχρονα που αξιολογώ την κατάσταση, υποκειμενικός φυσικά τρόπος, και ο τρόπος με τον οποίο αφού αξιολογήσουμε την κατάσταση διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα. Αυτά που μας κοστίζουν στο στρες είναι τα συναισθήματα. Σε αυτή τη συναλλαγή, συνδιαλλαγή υπάρχει ένα καθοριστικός, ένας καθοριστικός παράγοντας, η κοινωνική υποστήριξη. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι αν έχετε κοινωνική στήριξη υψηλή ποιότητας, η ικανότητά σας να απορροφήσετε το στρες είναι πολύ υψηλότερη. Ε, και αυτό είναι και πολύ σημαντικότερο για την επιχείρηση. Επίσης έχουμε τις συνέπειες, τις συνέπειες του στρες, γνωρίζουμε ότι είναι παράγοντας κινδύνου για την υγεία. Έχουμε το στρες από μόνο του σήμερα δεν θεωρείται ασθένεια, αλλά παράγοντας κινδύνου όπως η χολυστερίνη. Χολυστερίνη έχουμε όλοι, από ένα κατόφλιο και πάνω ε, διατρέχουμε κίνδυνο εφόσον το ύψος της χολυστερίνης είναι υπερβολικά υψηλό αλλά από μόνη τη χολυστερίνη δεν είναι ασθένεια. Αποτελεί κίνδυνο για την υγεία με τι συνέπειε που γνωρίζουμε, την αίσθηση ευημερία και τον κίνδυνο ε, διαφόρων ασθενειών λόγω του στρες. Γιατί σας δείχνω αυτό το μοντέλο, διότι όπως βλέπετε ο μεγάλος κίνδυνος που έχουμε, ειδικότερα στην περίπτωση του επαγγελματικού στρες, είναι ότι μετράμε το άτομο πώς είμαστε, πόσο στρεσαρισμένοι είμαστε, στη συνέχεια υπολογίζουμε τα στοιχεία, τους παράγοντες ε, πρόβλεψης, ε, τους συντελεστές ε, δηλαδή του στρες και κάνουμε ένα συσχετισμό μεταξύ των συντελεστών αυτών και της κατάστασης του ατόμου. Εξορισμό, όπως βλέπετε, πρόκειται για ένα μοντέλο λανθασμένο, διότι στο πλαίσιο της επαγγελματική ζωής δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις υπόλοιπε παραμέτρους που είναι εξίσου σημαντικές για το επίπεδο στρες του ατόμου. Αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να μετρήσουμε το τεστ, να το αξιολογήσουμε μέσω της κατάστασης των ατόμων, ώστε να γνωρίζουμε ποιος κινδυνεύει, ποιος υποφέρει πραγματικά και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν που υποφέρει. Ωστόσο θα πρέπει επίσης να προσέχουμε τις συνδέσεις που κάνουμε λίγο γρήγορα, ότι το, η εργασία για παράδειγμα προκαλεί στρες στον άνθρωπο ή ότι η ζωή η σημερινή ε, ε, δημιουργεί τέτοιο στρες. θα σας προκαλέσω λίγο και θα επιμείνω σε κάτι που μου φαίνεται πολύ ουσιαστικό για το στρες. Το στρες αντιστοιχεί στο κόστος προσαρμογής στην πίεση. Ε, ε, την έννοια της προσαρμοστικότητας. Τι είναι το στρες, πόσο μου κοστίζει το να προσαρμοστώ σε μια νέα κατάσταση δυσχερή, σε περιορισμούς και σε πιέσεις που υποχρεούμε να αντιμετωπίσω πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το ζήτημα της προσαρμοστικότητας που μας αφορά όλους και που είναι ένα ζήτημα όχι μόνο επαγγελματικό αλλά και ζωής, αυτή η προσαρμοστικότητα σχετίζεται άμεσα με μια εκπαίδευση που έχουμε λάβει όλοι μας ε, στην προσαρμογή. την ημέρα που σταματάμε να προσαρμοζόμαστε, που σταματάμε να δίνουμε κίνητρα στα άτομα για να προσαρμοστούν, χάνουν την ικανότητα προσαρμογής τους. Αυτό τι σημαίνει ότι σε μια επιχείρηση όπου έχουμε αφήσει τους ανθρώπους χωρίς να τους τρεσάρουμε καθόλου, λέγοντας τους συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε, μην αλλάξετε τίποτα για πολλά χρόνια. Αυτά τα άτομα χάνουν κάθε ικανότητα προσαρμογής και ένα πολύ μικρό στρες για αυτούς αποτελεί σημαντικό γεγονός και απαιτείται τεράστια προσπάθεια για την προσαρμογή. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πολύ. Η ιδέα ότι δεν χρειάζεται να έχουμε στρες στην επιχείρηση, το μοντέλο δηλαδή της ε, συνταξιοδό, της, ε, της απόσυρσης μάλλον, της απόστασης όπου δεν έχουμε πλέον πιέσεις, όταν δεν έχουμε πλέον περιορισμούς και πιέσεις και δεν χρειάζεται να προσαρμοστούμε σε κάτι, πολύ γρήγορα χάνουμε τις ικανότητες προσαρμογή. Καθώς ζούμε σε έναν κόσμο όπου απαιτείται όλο και περισσότερη προσαρμογή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία αποσταθεροποιούμαστε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Στην επόμενη διαφάνεια επιμένω στο γεγονός ότι το στρες είναι ένα υποκειμενικό φαινόμενο. Δεν είναι, φυσικά μπορούμε να το μετρήσουμε, είναι μετρήσιμο. Δεν είναι η πίεση, είναι πώς αντιλαμβάνομαι εγώ την πίεση. Αυτό είναι το στρες. Αυτή η αντίληψη είναι συναισθηματική τι είναι το στρες, μία ζυγαριά ουσιαστικά, μία ισορροπία μεταξύ του πώς εγώ αντιλαμβάνομαι την πίεση και πώς αντιλαμβάνομαι τις ικανότητες αντίδρασής μου. Είμαι ικανός να αντιδράσω κατά τη συναλλαγή που σας έδειξα προηγουμένως. Αυτό συμβαίνει μέσα στον καθένα μας. Είμαι ικανός να αντιδράσω και κατά κάποιον τρόπο ε, σε αυτή την πίεση που υφίσταμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα στις επιχειρήσεις έχουμε καταργήσει με φαινόμενα τα οποία θα προσπαθήσω να σας περιγράψω την αντίληψη που έχουν οι μισθωτοί όσον αφορά την ικανότητά τους να αντιδράσουν. Στο επόμενο στάδιο δηλαδή έχουμε, τοποθετήσει, στάδιο, έχουμε τοποθετήσει τους ε, ε υπαλλήλου σε μια κατάσταση θυματοποίηση όσον αφορά την κατάστασή του στην εργασία και όσο περισσότερο αισθάνονται θύματα, Όσο περισσότερο αισθάνεστε θύματα, τόσο περισσότερο αυξάνεται το στρες σας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε έναν φαύλο κύκλο, μέσα στον οποίο εγκαθίσταται ένα άτομο που έχει την αίσθηση ότι αποτελεί θύμα του συστήματος, ότι δεν μπορεί να αντιδράσει. Το άτομο σε αυτή την περίπτωση έχει μια αντίληψη του στρες πολύ ισχυρότερη. Το ζήτημα εκεί είναι μπορώ να αντιδράσω, να ρωτιέται κάποιο ε, στην πίεση. Αυτή λοιπόν η συστημική συνέπεια της θυματοποίησης και της, ε, άμβλησης του, και της ε, αύξησης του στρες. Πώς σχετίζεται αυτό με τις σχέσεις, εργασιακές σχέσεις. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, καθώς εργάζομαι σε διάφορες επιχειρήσεις παντός είδους, σε διεθνές επίπεδο και ε, στη χώρα μου φυσικά ε, παρατηρούμε σε ποιο βαθμό η υποβάθμιση της ε, σχέσης ε, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των μισθωτών αφενών και των επιχειρήσεων αφετέρου. Ο πρώτος λόγος φυσικά είναι η επικέντρωση των επιχειρήσεων σε οικονομικούς στόχους. Το γεγονός ότι έχουμε διευθυντές και μετόχους οι οποίοι ε, λειτουργούν μόνο με γνώμονα την αξία της επιχείρησης, ε, τα κέρδη της, τον τρόπο με τον οποίο θα έχουμε ε, βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των επενδύσεων και αυτό προκαλεί θυματοποίηση των συνεργατών και σήμερα με τις τελευταίες μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά τις σχέσεις των συνεργατών μέσα σε επιχειρήσεις παρατηρούμε ότι το 65% στη Γαλλία, βάσει μιας γαλλικής μελέτης, 65% των συνεργατών θεωρούν ότι το συμφέρον τους δεν είναι το ίδιο με αυτό των διευθυντών τους. Αυτό τι σημαίνει ότι κάθε φορά που ένα διευθυντή μια επιχείρηση λαμβάνει μια απόφαση, ο συνεργάτη πιστεύει ότι ο διευθυντή λαμβάνει την απόφαση για τον εαυτό του, για τα δικά του συμφέροντα και όχι για την επιχείρηση. Όσον αφορά αυτό, αυτή η αίσθηση θυματοποίηση είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θεωρώ ότι είμαι θύμα ενό χρηματοοικονομικού συστήματος στο οποίο δεν μπορώ να παρέμβω και δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να το υποστώ. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται οι επιχειρήσεις και η οργάνωσή του Σήμερα τα ε, δυνατά σημεία της, ε, των οργανώσεων ε, θα σας αναφέρω ουσιαστικά τρία σημαντικά σημεία για τις οργανώσεις. Το πρώτο είναι η εξατομίκευση της απόδοσης. Με πολύ έντονο τρόπο αυτό σημαίνει ότι έχουμε πιέσει ώστε καθοριστικό στην αξιολόγηση των εργαζομένων να είναι ε, το άτομο. Να απομονώσουμε δηλαδή απολύτως το άτομο στην επιχείρηση και να μην έχουμε πλέον ένα ε, τον κοινωνικό διάλογο και την ποιότητά του. Δεν λειτουργούμε πλέον ως συλλογική ομάδα, αλλά ατομικά. Ε, έτσι ξαφνικά ο κοινωνικός διάλογος δεν μας αφορά. Το μόνο που με αφορά είμαι εγώ ενώπιον της επιχείρησης. Αυτή η εξατομήκευση της αποδόσης ε, θέτει το άτομο σε μία ε, απώλεια ισορροπίας, διότι μόνος το έχει να αντιμετωπίσει την επιχείρηση. Η δεύτερη μεγάλη τάση που βλέπουμε σε όλες ε, στις, ε, στις ε, επιχειρήσεις είναι οι διεργασίες, η επαναπροσαρμογή θα λέγαμε των επιχειρήσεων. Ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μπορέσει να δούμε και που ειδικά στη Γαλλία προκαλεί, όλα τα δράματα που ε, έχουμε μάθει, όλε οι αυτοκτονίε που έχουμε ακούσει σε διάφορε επιχειρήσει ε, και βάσει των οποίων έχουν γίνει πολλέ αναλύσει. Το process αυτή, η διαργασία, μία σειρά από κανόνε που επιβάλλονται σε όλου, έχει αντικαταστήσει τη διαχείριση. Κανένα δεν έχει πλέον περιθώριο δράση, όλα προαποφασίζονται στο πλαίσιο διεργασιών, διαδικασιών. Φυσικά, έτσι λοιπόν οι διευθυντές και οι υπάλληλοι είναι εκτελεστικά όργανα. Τα εκτελεστικά η ύπαρξη αυτή εκτελεστικών οργάνων δημιουργεί την αίσθηση θυματοποίησης και ότι δεν υπάρχουν μέσα αντίδραση και φυσικά αυτό αυξάνει το επίπεδο του στρες. Επίσης, εξαιτίας της εξατομίκευση ε, υπάρχει η κατάργηση αυτού που ονομάζουμε κοινωνική στήριξη. Αυτό θα μπορούσε να απορροφήσει το στρες ε, η κοινωνική υποστήριξη σημαίνει το σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ όταν χρειάζεται να μιλήσω για κάτι, όταν θέλω να ζητήσω βοήθεια, όταν θέλω να συζητήσω κάτι. Το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένες διεργασίες για τις ε, διάφορες λειτουργίες, ε, αυτό προκαλεί κατάργηση, ουσιαστικά λέμε στου ανθρώπου ότι πρέπει να κάνουν μόνο κάτι συγκεκριμένο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούν και αυτό καταργεί την υποστήριξη από τους ε, δίπλα, από, τους, ε, από τη διαχείριση, από τη διοίκηση, από τους συναδέλφους. Ένα τρίτο σημείο πολύ σημαντικό που εξηγεί αυτές τις ε, σχέσεις είναι αυτή η απόσταση μεταξύ της ε, προσδοκίας ε, για πρόοδο που είχαν οι προηγούμενες γενιές, ε, προσδοκία για προ... ιεραρχική πρόοδο, για προαγωγή ουσιαστικά, το οποίο δημιουργεί μια αίσθηση δυσχερίας και οι δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι προς το τέλος της διαδρομίας τους. Με λίγα λόγια, τι θα μπορούσε, πώς θα μπορούσαμε να μελετήσουμε και να σκεφτούμε νομίζω ότι το στρες δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε από τη στιγμή που μπορούμε να το μετρήσουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να μπορούμε να καταμετρήσουμε, να υπολογίσουμε το στρες, το επίπεδο του στρες του πληθυσμού στο χώρο εργασίας, επειδή αυτό αποτελεί δίκτυ, το σημαντικότερο πιστεύω δίκτυ, που επιτρέπει να παρακολουθούμε χονδρικά την κατάσταση των εργαζομένων. Σήμερα η κίνδυνη υγείας ε, στην ε, εργασία είναι ψυχολογική κυρίως. Έτσι έχουμε περάσει τα όρια που υπήρχαν προηγουμένων. Τα όρια του στρες δεν είναι ορατά από κανέναν και ε, εντείνονται όλο και περισσότερο. Όταν μιλούσαμε για σωματικά όρια μπορούσαμε να δούμε τα όρια αυτά. Υπήρχαν σωματικά συγκεκριμένα όρια. Σήμερα στα ψυχολογικά όρια δεν έχουμε ορατότητα. Δεν μπορούμε να δούμε ποια είναι ακριβώς τα όρια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να μετρήσουμε το στρες με δύο θεμελιώδεις παράγοντες. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ατομικό από το συλλογικό. Υπάρχουν ζητήματα ατομικού στρες που πρέπει να αντιμετωπιστούν ατομικά χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε όλες τις πιέσεις. Υπάρχουν προβλήματα συλλογικού στρες στην επιχείρηση και εκεί πρέπει να αναρωτηθούμε τι πίεση υφίστανται οι συνεργάτες και να ελαττώσουμε αυτή την πίεση. Υπάρχει σύγχυση μεταξύ αυτών των διαστάσεων, πιστεύω πολύ σημαντική. Ε, επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι σε μια επιχείρηση έχετε πάντοτε ένα κομμάτι των εργαζομένων που δεν πάνε καλά και ένα άλλο κομμάτι που αισθάνεται καλά. Ε, το να ελέγχουμε το στρες καθολικά για όλους συνήθως είναι αναποτελεσματικό. Πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε το στρες για όσους δεν αισθάνονται καλά. Τέλος όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, μερικές προτάσεις που θα μπορούσαμε φυσικά να αναπτύξουμε και άλλες όπως βλέπετε στις εντάσεις μεταξύ των ενδιαφορομένων πρέπει να ξαναδώσουμε στην επιχείρηση με νομικά και δημοσιονομικά μέσα τη δυνατότητα να έχουμε να λαμβάνουμε κάποια σχόλια από τις επιχειρήσεις στα επιχειρηματικά θέματα. Μπορούμε για παράδειγμα να θα την εξαγορά με μετοχών. Κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, οι συνεργάτες καταλαβαίνουν ότι προσπαθεί η επιχείρηση να ευνοήσει τον μέτοχο, να βγάλει κέρδη και θέτουμε λοιπόν την επιχείρηση σε ένα κίνδυνο βιώσιμης ανάπτυξης διότι όλα εξαρτώνται από την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν κάνει πιο τους διευθύντες και τους μετόχους εις βάρος της επιχείρησης. Έτσι θυματοποιούνται οι άνθρωποι περισσότερο και αυξάνεται το στρες. Ε, το ζήτημα της αμοιβή φυσικά των ε, διευθυντικών στελεχών αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Δίνει την ε, εντύπωση ενός τεράστιου χάσματος, ε, αβυσαλέου χάσματος μεταξύ ανθρώπων ενός συγκεκριμένου επίπεδου εισοδημάτων και άλλων που κερδίζουν πολλά περισσότερα έχουν την αίσθηση της αδικίας. Επίσης το ζήτημα της φορολογίας. Ε, σήμερα όπως γνωρίζετε το φορολογικό σύστημα σήμερα φορολογεί ε, ευνοεί κατά κάποιο τρόπο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ε, δεν υπάρχουν διακρίσεις σε αυτό το επίπεδο όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας. Μου φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε να αντισταθμίσουμε την ατομική πτυχή της απόδοσης με τη συλλογική πτυχή ώστε να αναδιορθώσουμε το κοινωνικό περιβάλλον των συνεργατών ώστε να αισθάνονται ότι περιβάλλονται από ένα φιλικό ε, από φιλικές συνθήκες. Οι σταδιοδρομίε σήμερα μεταβάλλονται πολύ πιο γρήγορα, έτσι λοιπόν υπάρχει ανάγκη να γίνονται πιο τακτικοί απολογισμοί Τη εξέλιξη της ε, σταδιοδρομία. Οι σταδιοδρομίε είναι πολύ πιο μακροχρόνιες και έτσι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι λαχανιασμένοι στην εργασία. Ε, χρειάζονται ε, έξι μήνε μήνες ή ένα χρόνο, καμιά φορά παίρνουν οι άνθρωποι μακριά από την εργασία τους. Ε, υπάρχει ένα παράδοξο, οι άνθρωποι στο τέλο τη διαδρομίας του κερδίζουν περισσότερα χρήματα και είναι λιγότερο παραγωγικοί. Μου φαίνεται προφανέ ότι θα χρειαστεί να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις περιόδους τέλους σταδιοδρομίας για φυσικά εντάξει λιγότερη παραγωγικότητα αλλά να μπορεί να ευνοήσει τη λειτουργία της επιχείρησης με λιγότερο υψηλές αμοιβέ στο τέλος της σταδιοδρομίας. Για να συμπεράνω, για να φτάσουμε στα συμπεράσματα, προσοχή να μην είμαστε υπερβολικά ιδεολόγοι και να μην υπεραπλουστεύουμε την ε, σχεσιακή διάσταση του στρες και να μην κρυβόμαστε πίσω από το στρες ως μιας τεχνικής έννοιας. Πρέπει να καταλάβουμε το στρες στην εργασία είναι ένα ζήτημα πολύ πρόσφατο όπου οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν καν πανεπιστημιακές έδρες για αυτό το ζήτημα. Έχουμε λοιπόν ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα. Έχουμε έλλειψη επιστημονικών δεδομένων. Ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσατε να προτείνετε να υπάρχουν πανεπιστημιακές έδρες για το στρες στο χώρο εργασία. Πρόκειται για το θέμα που τίθεται σήμερα όσον αφορά την ε, υγεία στο χώρο εργασία. Αυτά είχα να σα πω. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Nous avions euh, avant-hier un échange avec Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή της Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας είπε ότι στο θέμα της απασχόλησης θα πρέπει να έχουμε δείκτες και δεδομένα, αξιόπιστα δεδομένα, μετά από παρατήρηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιδράσουμε επί της συζήτησης, ιδιαίτερα στους υπεύθυνου των χρηματοοικονομικών. Να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Η Καρίν Μαντελή έχει το λόγο και μετά ο, κύριο, ο αντιπρόεδρος μας, ο κύριος Τόμας Μαν. Η κυρία Ντελή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Νομίζω ότι σήμερα όταν μιλάμε για στρες θα πρέπει να αναλύσουμε τους παράγοντες ε, που επισύρουν το στρες και πώς μπορούμε να δράσουμε για να προλάβουμε, για να μειώσουμε το στρες. Άρα όλες οι προληπτικές ε, πολιτικές είναι αναγκαίες. Δεν επιμείνετε σε αυτό, θα ήθελα να επανέλθετε. Επίσης θεωρούμε ότι το στρες επηρεάζει στην απόδοση και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η οργάνωση εργασίας, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την εργασία, διότι η διαχείριση έχει αλλάξει πλέον. Και σήμερα έχουμε τρόπους που επιβάλλονται χωρίς κοινωνικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οπωσδήποτε αυτό επηρεάζει και την συλλογική αποδοτικότητα και την ατομική. Μιλήσατε. Euh, Για πανεπιστημιακές έδρες, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι όχι μόνο να τα τονίσουμε ακαδημαϊκά όλα αυτά, αλλά να τα δούμε in situ, στην εργασία. και να γίνει ένα είδος κατάρτισης για το πώς μπορεί κανείς να διαχειρίζεται το στρες. Δηλαδή να λάβουμε αυτή τη θεματική ενότητα και να την αναπτύξουμε. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή στρατηγική, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι σκέφτεστε. Πιστεύετε ότι το στρες στο χώρο εργασίας λαμβάνεται παρκώ υπόψη στις δημόσιες ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, νομίζετε ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας των Ευρωπαϊκών Εταίρων για το στρες έχει λειτουργήσει, δεν έχει λειτουργήσει, πού πρέπει να προχωρήσουμε ως προς τη στρατηγική αυτή και τέλος. Πιστεύετε ότι η νομοθεσία έχει θετικό αντίκτυπο ως προς το στρες στην εργασία θα πρέπει να έχουμε μια οδηγία για το στρες στην εργασία που να εμπνέεται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων. Και σήμερα χρειαζόμαστε πράγματι κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να, να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η οδηγία, αλλά εσείς ως εμπειρογνώμων θεωρείτε ότι πραγματικά πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Ωραία. Ανεβαίνει το στρες. Θα ήθελα λοιπόν οι συνάδελφοι που παρεμβαίνουν να είναι πιο σύντομοι. Ο κύριος Τόμας Μαν, Μωρέ, Χάντελ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο. Φαίνεται πως όχι. Κλείνει ο κατάλογος και δίνω το λόγο στον κύριο Τόμας Μαν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα όλα αυτά τα στοιχεία από τον κύριο Αλμπέρ. Έχετε μια θαυμάσια ευκαιρία να γνωρίσετε κόσμο, ο οποίος μπορεί να χειριστεί θαυμάσια αυτό το στρες. Είναι όλοι εδώ οι παρόντες, οι οποίοι κάθε μέρα ε, περνάνε, όπως λέμε, ζωή και κότα. Ε, όλοι οι ευρωβουλευτές έρχονται εδώ χαρούμενοι το πρωί, τραγουδώντας, ε, περνάνε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα, άνετα, ε, παραχαϊδεύουν τους βοηθούς τους και είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, χαρούμενοι και ξεκούραστοι. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι ένας τέτοιος κόσμος δεν υπάρχει. Τώρα, πέραν της πολιτικής, αυτά που έχω μάθει στον εργασιακό χώρο, το, το πιο σημαντικό πράγμα για να ξεπεράσουμε αυτό το στρες ή για να το αντιμετωπίσουμε, είναι ότι χρειαζόμαστε μια σωστή αξιολόγηση. Εσύ ως εργαζόμενος, παραδείγματος χάρη, δεν αναγνωρίζεις, δεν ξέρεις ακριβώς τι σου συμβαίνει. Για να μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και να χειριστούμε αυτό το φαινόμενο του στρες, χρειάζεται μια σωστή αξιολόγηση, μια αναγνώριση του φαινομένου. Πολλέ φορές οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι θα με κρίνουν αρνητικά, ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις εάν το ομολογήσω. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πώς γίνεται η αξιολόγηση ενός εργαζόμενου και από τον προϊστάμενο και από τους υφιστάμενους και ότι πολλές φορές τα φαινόμενα ερμηνεύονται με εντελώ διαφορετικά κριτήρια, με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Καμιά φορά ε, λες το παράπονο σου, το πρόβλημά σου και ο, αυτός που σε ακούει σου λέει σταμάτε επιτέλους δεν μπορώ να σε ακούω άλλο. Ε, τι είναι αυτά που μου λες. Πρέπει λοιπόν αυτό το, αυτή η δυνατότητα, αυτό το θάρρος που χρειάζεται να σταθείς ενώπιον των άλλων και του αυτού σου και να ομολογήσεις το πρόβλημά σου. Το άλλο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος ένα χώρο δημιουργικότητας. Δηλαδή χρειάζεται ένας ε, ατομικός χώρος ο οποίος δεν ανήκει στους άλλους, ε, όπου δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος μέσα να μπορέσει κανείς να εργαστεί ε, και με άλλους συνεργάτες και σε ομάδες και να μπορεί να ομολογήσει την αλήθεια στους άλλους και να πει σε κάποιον ότι αυτό που έκανες δεν μ' άρεσε ή αυτό που μου δείχνεις εδώ δεν είναι καλό. Επίσης, η πίεση συνεργάζεσαι και το Σαββατοκύριακο. Εμείς ε, κάναμε διαφορετική οργάνωση. Ε, κάναμε ένα brainstorming με τους συνεργάτες όπου όλοι παρουσίαζαν τις ιδέες τους και πολλοί εργαζόμενοι μας είπαν ότι δεν χρειάζεται να φτιάξουμε έναν ωραίο χώρο, εικονικά, ιδανικό χώρο, τουλάχιστον να έχουμε μερικά δέντρα να βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να είναι όλα ιδανικά στον περιβάλλοντα χώρο. Ακούσαμε λοιπόν αυτές τις ιδέες και επίσης προσπαθήσαμε να αναθέσουμε σε κάποιον να ασχολείται με το θέμα αυτό του στρες. Και ε, δεν ήταν ένας εμπειρογνώμων ή ένας ειδικό, αλλά ήταν κάποιο άτομο το οποίο επιλέγαμε κάθε φορά, που ήταν μια πάρα πολύ σωστή επιλογή, διότι ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο μπορούσε κάποιος να πάει και να του εκφράσει το, το στρες του, να του πει τι γίνεται στην καθημερινή του ζωή και πιστεύω ότι αυτό ήταν μια καλή ιδέα. Ε, μπορέσαμε κάπως να διαχειριστούμε και να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι διοργανώσατε αυτή την ακρόση που είναι άκρος ενδιαφέρουσα σήμερα το πρωί και θα ήθελα να έχουμε τα έγγραφα. Όπως είπε η Καρή Μαντέλη για την πρόληψη του άγχους, δεν μιλήσατε κύριε, μάλλον είπατε ότι χρειαζόμαστε μισθούς προσαρμόσιμους αλλά δεν μιλήσατε για την κατάρτιση, διότι στην αρχική κατάρτιση θα ήταν άκρος ενδιαφέρον ήδη από το σχολείο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα προσαρμοστικότητας. Ο Τόμας Μαν το ανέφερε αυτό. Θα πρέπει να το δούμε στις επιχειρήσεις, αλλά από την παιδική ηλικία το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι πολύ δεσμευτικό και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της προσαρμοστικότητας. Το, πρώτο, το δεύτερο θέμα είναι το σε αυτόν. Ο Τόμας Μαν το είπε για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να ξέρουμε πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε, πώς μας κρίνουν. Or, on est dans un monde extrêmement cloisonné. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ζούμε σε έναν πολυμηνυματικό κόσμο. Et euh, la dimension du regard ε, θα πρέπει λοιπόν μέσα σε αυτόν τον κόσμο να ξέρουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη διάσταση του γνώθησε αυτόν. Το τρίτο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι ότι όπως είπατε το άγχος είναι ατομικό και συλλογικό και δεν είχαμε αυτή την ε, συνολική προσέγγιση. Στον ε, κοινωνικό λοιπόν διάλογο βλέπουμε ότι σε επίπεδο επιχειρήσεων έχουμε χάσει τον αντίκτυπο των συνδικάτων και ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνολική γνώση της επιχείρησης. Δεν καταβάλουμε το αντίτιμο σε ατομικό επίπεδο του γεγονότος ότι η παγκόσμια οργάνωση της ε, επιχείρησης έχει κάπως ξεφύγει. Πριν περάσουμε στο στρες της ψηφοφορίας, ο ε. Τόμας Χέντελ έχει το λόγο. Ε. Thomas Mann hat, äh, Ο Τόμας Μαν περιέγραψε πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία συμβαίνουν σε πολλές επιχειρήσεις και πώς αντιμετωπίζουν το καθημερινό στρες. Τον υποστηρίζω σε αυτά που είπα και συμφωνώ. φοβούμε όμως ότι υπάρχει ένα, το στρες που, για το οποίο συζητάμε είναι ένα συστημικό στοιχείο της ε, ενσωματωμένο στην καθημερινή δουλειά, στο καθημερινό περιβάλλον. Ένας μάνατζερ, ας πούμε, μιας μεγάλης εταιρείας της Intel εδώ και 15 χρόνια έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Μόνο η παρανοϊκή θα επιβιώσει». Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο μάνατζερ έγραψε ότι ο φόβος είναι το, η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη για την, ε, το μεγαλύτερο έναυσμα ε, της προς εργασία. Δηλαδή, αν οι εργαζόμενοι ζουν υπό συνεχή φόβο, είναι το, ο καλύτερος τρόπος να δουλεύουν. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι τεράστιες επιχειρήσεις και αυτός ο τρόπος του management στηρίζεται στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεχούς φόβου. Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι το 30% των Ευρωπαίων πολιτών πάσχει από ψυχικό, ψυχικό στρες ή διανοητικές ε, ασθένειες. Ε, επί λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή τη πρόταση οδηγία, πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με διαφορετικό τρόπο πλέον. Αλλά ένα στοιχείο λείπει από τη μελέτη σα. Στη Siemens στη Γερμανία είδα ότι το δόγμα μιας μεγάλης εταιρείας είναι να λέει ε, να λένε οι μάνατζερ στους εργαζόμενους ότι τους μισθούς σου ε, δεν τους πληρώνει η εταιρεία, τους πληρώνουν οι πελάτες. Ε, το, οποίο παρουσιάζουν δηλαδή μία εικόνα ότι η εταιρεία άγεται και φέρεται από εξωτερικά στοιχεία και ότι δεν είναι σε θέση μέσα στο περιβάλλον εργασίας να λαμβάνει τις αποφάσεις που πρέπει, δημιουργώντας ένα ακόμα στοιχείο, ένα ακόμα επίπεδο φόβου Ευχαριστώ πολύ. Αλεχάνδρο Σέρκος. Και μετά ο Ρίτσαρντ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Πρώτα να ευχαριστήσω γιατί ήταν μια εισήγηση πολύ ενδιαφέρουσα. Δεύτερον, για να κάνω δύο ερωτήσεις για δύο θέματα που είναι λιγότερο σαφή αυτά τα δύο θέματα. Είναι πολύ σαφής η προσπάθεια να παρουσιαστεί να παρουσιαστούν οι επιπτώσεις του στρες του άγχους σε μια κατάσταση επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ας την αποκαλέσουμε, στον εργατικό εργασιακό τομέα ή επαγγελματικό τομέα που βρίσκονται ακριβώς στην αιχμή όσον αφορά την παραγωγή της συνδιαλλαγής. Αλλά δεν είναι σαφές τι γίνεται με εκατομμύρια ανθρώπους που κάνουν επαναληπτική δουλειά, μονότονη δουλειά, που δεν είναι και τόσο υγιεινή και ήμουνα εισηγητή για τον χρόνο εργασία. Εν τέλει θα ήθελα να ξέρω, ο υπερβολικός χρόνο εργασία, σε τέτοιου είδου εργαζόμενου, δεν έχει μια επίπτωση δημιουργία άγχου, δεν δημιουργεί στρες και είναι αυτό σοβαρό για τις επιπτώσεις ε, για τη δική τους προσωπική ζωή και προς την ίδια κατεύθυνση. Δεύτερη ερώτηση. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα της προσαρμογής είναι το κλειδί του προβλήματος του άγχους. Και βλέπουμε εδώ η προσαρμοστικότητα προάγεται για τους εργαζόμενους και για τις αλλαγές. Έχω μια αμφιβολία. Αυτό δεν, έχει, δεν είναι μια πραγματικότητα με δύο όψεις. Η προσαρμοστικότητα επίσης από την άλλη πλευρά των επιχειρήσεων στις ανάγκες των εργαζομένων. Και αυτό δεν αποτελεί ένα στοιχείο που πέρα από τη δημιουργία στρες για τους εργαζόμενους και μέσω των αλλαγών που δημιουργούνται οι ίδιες οι επιχειρήσεις στις αλλαγές να ξέρουν ότι δεν είναι μηχανές οι άνθρωποι και ότι πρέπει και εκείνες να κάνουν μια προσπάθεια προσαρμογής στις ουσιαστικές δυνατότητες απόδοσης των εργαζομένων. Είναι μονομερή προσαρμοστικότητα από πέρα των εργαζομένων μόνο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ είναι σαφές και ήθελα να πω ότι πάντα όταν βλέπουμε τον πίνακα ψηφοφορία, όταν εγώ βλέπω τον πίνακα ψηφοφορία, μου δημιουργείται άγχος στρε. Και όταν έχουμε την άσκηση, το εγχείρημα στην Επιτροπή μας για κάθε έκθεση να υπάρχουν 500 ή και παραπάνω τροπολογίες, πάλι άγχος, στρες δημιουργείται. Δεύτερον, δεν γνωρίζαμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ήδη ότι είναι τα συνδικάτα σε σχέση με τα τελευταία φράγματα που υπάρχουν ή αναχώματα προτού το αόρατο χέρι της αγοράς επιβληθεί και διαμορφώσει τα πάντα. Δεν είδαμε και είμαστε μάρτυρες πολλές φορές αυτού του γεγονότος. Δεν είμαι μέλος. Γιατί διαρωτώνται τόσο πολύ οι Γάλλοι για αυτά. Τα συνδικάτα απαλήφθηκαν ακόμα και στις χώρες όπου είχαν μεγάλη εξουσία στο παρελθόν, μεγάλη δύναμη και επιρροή και για πολλούς λόγους. Και τρίτον, ελπίζω ότι το συμπέρασμα αυτών δεν θα είναι μια νέα οδηγία που θα συνταχθεί όσον αφορά τη στρατηγική από, την, από πλευράς Ευρώπης για την καταπολέμηση του στρες. Ευχαριστώ. la diversité existe. Υπάρχει διαφορετικότητα και αποκλήσεις και στη δική μας Επιτροπή και σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε σύντομα σε αυτές τις ερωτήσεις και θα σας ζητούσα να μας δώσετε την... και το PowerPoint, την παρουσίασή σας. Η Καρή Μαντέλη ρώτησε κατά πόσο το άγχος λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Πολύ πρόσφατα γίνεται αυτό βλέπουμε ότι πρόκειται για εξωγενείς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη και με βάση και την πίεση της κοινή γνώμης λήφθη υπόψη. Δηλαδή στη France Telecom μετά τις αυτοκτονίες είδαμε ότι πρέπει το άγχος να αρχίσουμε το να τον λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί πριν δεν συνέβαιναν και πολλά. Σήμερα λαμβάνεται υπόψη ε, αλλά περιθωριακά, δηλαδή ως επιφαινόμενο. Γίνονται δύο-τρεις συμφωνίες και δεν τίθεται θέμα ουσίας. Δηλαδή να δούμε ποιε ποιες είναι οι πληθυσμιακές κατηγορίες που πλήττονται, ποιες δεν τα καταφέρουν στις, στην προσαρμογή ποιες είναι οι οργανωτικές δεσμεύσεις, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις κατηγορίες. Καταβάλουμε ε, το, την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια, περιφερειακά. Τώρα πρέπει να νομοθετήσουμε. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί δεν υπάρχει καθολική λύση και επίσης ε, ε, δεν μπορεί ο νόμος να αντιμετωπίσει το καθολικό αυτό φαινόμενο. Εάν όλοι προβαίνουμε σε μετρήσεις, μετά θα πρέπει να λογοδοτήσουμε. Τη στιγμή που δεν έχουμε μετρήσει τίποτα, τη στιγμή που δεν απαριθμούμε προβλήματα, δεν ξέρουμε την κατάσταση. Όταν τα απαριθμίσουμε, ε, όλους αυτούς τους παράγοντες και τους δείκτες. Αν έχουμε 30, ε, από 35-30 πάμε καλύτερα. Αν από 30-35 το αντίθετο. Ο Τόμας Μαν είπε, έθιξε ένα κέριο ζήτημα. Δηλαδή ποιο είναι το διακύβευμα θα πρέπει σε τακτά χρονικά ε, διαστήματα να βγαίνουμε από την ε, ε, ανάπαυσή μας και να δούμε κατά πόσο αναπαράγονται συγκεκριμένες συμπεριφορές. Αυτή είναι, αυτό αποτελεί και τη γύρανση. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Μπορεί κανείς να θεωρείται γέρος στα 40 χρόνια και να μην είναι στα 80-90. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι η δυνατότητα να αμφιβάλλει κανείς και να έχει άλλους τρόπους συμπεριφοράς, να προσαρμόσεται, διότι ε, απότοχο του γύρατος είναι κανείς να μην λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον του. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Μωρέν για την αρχική κατάρτιση, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ε, πολύ σημαντικό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η ανάπτυξη των παιδιών μας είναι καθαρά πνευματική και ξέρουμε ότι η επιτυχία τους εξαρτάται από την συναισθηματική ευφία. Για ένα παιδί 10 ετών δεν έχει σημασία το IQ του, αλλά η συναισθηματική του ευφία. Και αυτή δεν αναπτύσσεται στο σχολείο. Είναι ένα μείζον ζήτημα. Γιατί βλέπουμε ότι ε, αναπτύσσεται το παιδί πνευματικά σαν να ήταν και το μόνο σημαντικό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η συναισθηματική ευφία. Ως προς τη διαχείριση μέσω τρομοκρατίας, συμφωνώ ότι αυτή η τάση αναπτύχθηκε. Όσο υπάρχει διαχείριση με τρομοκρατία, τότε έχουμε δημίους. Άρα οι δήμοι δεν ε, δημιουργούν προστιθέμενη αξία, αλλά στην ουσία υπόσχονται στον πελάτη μία χαμηλή τιμή. Δεν είναι το low cost το μέλλον της Ευρώπης, αλλά η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η δυνατότητα δημιουργίας αξιών. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω τρομοκρατία, διότι αν έχουμε διαχείριση μέσω τρομοκρατία, τότε κανένας δεν αναλαμβάνει κίνδυνο. Και αυτό που έχει σημασία είναι πέρα από το θέμα του άγχους να δούμε και το μέλλον της επιχείρησης, το οποίο διακυβεύεται. και ως προς τις ε, δεινές, τη δυνότητα της εργασίας μπορώ να μιλήσουμε για ωράρια, για μέσα μεταφοράς, για εργονομικές παραμέτρους που έχουν μελετηθεί και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τις απτές επιπτώσεις που όλα αυτά μπορεί να έχουν επί του άγχους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό ε, αυτή τη στιγμή για την Επιτροπή μας. Βρισκόμαστε σε ε, ανεξερεύνητο ε, εδάφη αυτή τη στιγμή για εμάς. Αυτή η εξέλιξη, η εξατομίκευση των επιχειρησιακών δομών, οι σύγχρονες μορφές του καπιταλισμού και οι συνέπειες του για την κατάσταση των απασχολούμενων ε, πιστεύω για τη δική μας επιτροπή αν θέλουμε να είμαστε πεφωτισμένοι νομοθέτες είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε και αυτή την προσέγγιση κύριε Καρή Μαντελή πιστεύω έχει ήδη βρει κάποια στοιχεία για να μπορέσει να εμπλουτίσει την έκθεσή της θα κατανέμουμε όλες τις πληροφορίες που μας δώσετε στο σύνολο των συναδέλφων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 12 και στην πρώτη ψηφοφορία που αφορά την έκθεση του κυρίου Φρέντερικ Νταρντέν ε, που αφορά την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βλέποντας τις 35 ε, σελίδες που έχουμε για την ψηφοφορία θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα. Η κυρία Εσάγια, στα πρακτικά της συνάντησης δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν ε, σκόπο να λεχθεί ότι είχαμε μόνο στα γαλλικά τις τροπολογίες συμβιβασμού. Θα ήθελα να, να καταγραφεί στα πρακτικά. Θα γίνει, θα γίνει και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι άκρος απογοητευτικό, δείκτης απογοήτευσης και αγχογόνος παράγων. Δυστυχώς για τις τροπολογίες συμβιβασμού αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Δεν τις έχει κανείς στη μητρική του. Όλοι έχετε την κάρτα σας. Λοιπόν, αρχίζουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τον τίτλο, μία τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται συμβαστική α, που υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, παράγραφος ε, 1 υπέρ κατά απορρίπτεται, 154 υπέρ κατά αποχές απο, εγκρίνεται, 155 του κ. Νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β από 5 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 παράγραφος Μπορούμε να τις δούμε σε Λίβδιν. Ωραία. 30, 13, 14, 15 και 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Παράγραφο 1. Τροπολογία G. 5 πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 2 σε 5 πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Μετά την παράγραφο 2, 1 της Επιτροπής ΦΑΜ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 Χέλμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 173 Όμιν Ράιτεν και άλλων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά τη 175 ε, των ιδίων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Δύο τροπολογίες ε, διαγραφής 176-177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβασμός Δέλτα. Πέντε πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. 184 Χέλμερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ε, 5 πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. F είναι συμβατός ο συμβιβασμός με προσθήκη προφορική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμο ε, ζ Ζ5 ομάδων στην παράγραφο 5 με προφορική προσθήκη υπέρ κατά απόχέ ε, εγκρίνεται. Παράγραφο 6 Α 5 πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6 199 Καρή Μαντέλη και άλλων υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 200 του εισηγήτη υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6 πάλι 202 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 203 του ιδίου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. Επί του τίτλου της παραγράφου 7 προφορική του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 7 υπάρχει μια τροποποίηση μου λένε. Δεν υπάρχει προφορική ή λοιπόν πέντε πολιτικών ομάδων τεσσάρων με συγχωρείτε, όπως προτάθηκε αρχικά υπέρ. Κατά αποχέ ε, εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 7, τροπολογία 208 του εισηγητή και άλλων υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 209 καταπίπτει, άρα ψηφίζουμε την πρόταση συνδυασμού Κ. Πέντε πολιτικών ομάδων υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 2.11 καταπίπτει. Φτάνουμε λοιπόν στην τροπολογία 2.15 του κυρίου Μπλό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 7 2.16 τροπολογία Καρή Μπαντελή υπέρ κατά Ήθελα να σας κάνω λίγο γυμναστική σήμερα και να αλλάξουμε ίσως ε, τις... Ε, ωραία, άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για την 2.15. Κατ' εξαίρεση έχω μία ε, κάρτα ψηφοφορίας, αλλά δεν λειτουργεί. Ah, Ακυρώνουμε λοιπόν και ξεκινάμε από την αρχή. Τα μηχανήματα φαίνεται ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν. Ε, έρχεται η ψηφοφορία. Γιατί το δικό μου ανάβει και του διπλανού μου. Ανάβει το διπλανό. Το μηχάνημά μου δεν λειτουργεί, έτσι δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε επαλήθευση. Ε, ε, ε. Λειτουργούν όσα είναι δίπλα μου όμως, όχι τα δικά μου. Εγώ ψηφίζω ναι και μου βγάζει όχι. Λοιπόν, θα το κάνουμε ως χείρος. Ποιος είναι υπέρ της 2.15. Υπέρ της 2.15. Υπέρ της 2.15. Σας είπα ότι είχα δίκιο, ε. Ποιος είναι κατά. Χρειάζεται πραγματικά να μετρήσουμε. Bon, allez. Mais bien sûr, monsieur. Et qui s'abstient apoches 17 17-25-2, l'amendement 215 de monsieur Philippe Boulange. 2-15, κύριε Φιλιμπουλόν, ζητώ συγγνώμη, δεν εγκρίθηκε όπως σας είχα πει ότι θα γινόταν. Ελπίζω ότι οι τεχνικοί μας θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των μηχανημάτων, γιατί εδώ έχουμε κάποιο μικρό προβληματάκι. Ε. Προσπαθούσαμε να αξιολογήσουμε την ικανότητά μας αντιμετώπιση του στρες. Το 2016, κυρία Καρύμαντέλη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, 2, 17, καταπίπτει, θέτω στη ψηφοφορία τη συμβαστική M της παραγράφου 8 με προφορική του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική L με προφορική τροπολογία υπέρ κα, υπέρ Qui est Κατά αποχές Εγκρίνεται. 217 Φτάνουμε στη 217. Συγγνώμη, 2.27. 2.17 το κάναμε. 2.27. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 2.28 της κυρίας Φιγκερέντο. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 2.29 του κυρίου Πουπάκη. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε παράγραφο 8.2.32 τσίμερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.33 τσίμερ πάλι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 2.34 της Κυριαντέλη και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.35 κύριο Πουπάκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.36 235 και pour le 200... 235 ποιος είναι υπέρ, κατά. On va, va, va, va voir si les machines marchent. Να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα, όχι δεν λειτουργούν. Ποιος είναι υπέρ της 235. Qui est contre Kata. Qui s'abstient apoches 25 25-21-0. 25-21-0. Εγκρίνεται 2-36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.37 του κ. Νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.38 του κ. Νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 8 ακόμη ε, στο 17 της Κουλτούρα ε, υπέρ κατά απορρίπτεται, 18 της ίδιας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9, συμβιβαστική 1 από 4 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε παράγραφο 10 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται της ίδιας Επιτροπής υπερκατά κατα 7 υπερκατά 2.48 καταπίπτει 2.49 ψηφίζουμε της κυρίας Αρκίν υπέρ 2.49 2.47 κατέπεσε qui est 247 υπέρ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 Qui Αποχές. 28-17 εγκρίνεται. 2.49 τη κυρία Αρκίν υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε Ποιο είναι υπέρ τη 2.49 υπέρ τη 2.49 Ε, τώρα είναι σαφές. Απορρίπτεται. 2.50 της κυρίας Λίν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.51 της κυρίας Ροντζούλη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.53 της κυρίας Ντέλη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Αποχές απορρίπτεται. Παραγραφός 5 της Επιτροπής Προπολογισμού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγραφός 10 συμβαστική όμικρον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 της Επιτροπής ΦΑΜ με προφορική υπέρ κατά εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 15 της ίδιας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 του κ. Ποπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 264 τσίμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 265 μπουλά πρώτο τμήμα ψηφίσουμε. χωρίς τις λέξεις would like to see national legislation και μέχρι can be terminated ποιος είναι υπέρ του τμήματο χωρίς αυτές τις λέξεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ποιος είναι υπέρ της προσθήκης κατά αποχές. Άρα γίνεται η προσθήκη 266 του εισηγητή και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 268 πουπάκης υπέρ κατά. Δεν είναι σαφές. Υπέρ της 268 του κυρίου Πουπάκη και άλλων. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11. 269 Χέλμερ υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβασμός π. Πέντε πολιτικών ομάδων με μία προφορική. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 11 ψηφίζουμε την πέντε της Επιτροπής Προπολογισμών. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 279 κοφεράτη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 280 ελ χέλμερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 281 κυρία Πλάμπ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 11, 284, κύρια Πλάμπ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 285, Νταρντέν και άλλων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12, συμβιβασμός Q. Πέντε πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ήταν τέσσερις πολιτικές ομάδες και όχι πέντε. Με μια προφορική. Μετά την παραγραφό 12, 293 τσίμερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 294 της κυρίας Πλάμπ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 295 και 96 είναι παρόμοιες. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτονται, αλλά θα επαληθεύσουμε. Γιατί ίσως δουλεύουν και τα μηχανήματά μας πλέον. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ας επαληθεύσουμε λοιπόν επί των 295-296. Ψηφίσατε. Μία ανθίσταται. Ένα μηχάνημα. Αν πείτε τι ψηφίσατε λοιπόν στο τέλος. Και τώρα λειτουργεί. Άρα είναι απολύτως απαραίτητη η τεχνική. Λοιπόν, ψηφίσατε αυτή τη φορά. Τρεις δεν ψήφισαν. Πέρασε. 46 ψήφισαν, 24 υπέρ, 22 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνονται λοιπόν 2,97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2,98 Λαμπέρ και άλλων υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νόμιζα ότι είχε απορριφθεί, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Alors. Ε, Μετά την παράγραφο 13, 299 Helmer για απόρριψη υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός R. Ορί. Euh, euh, Κύριε αυτός ο συμβιβασμός υποβλήθηκε από τέσσερις πολιτικές ομάδες. Εάν ε, θέλετε μπορώ να το αναφέρω ότι πρόκειται για την ΑΡ με μία προσθήκη που υποστηρίζεται από τους σοσιαλιστές, φιλελεύθερους, πρασίνους και γκουε. Ποιος είναι υπέρ της λοιπόν. αν Υπερψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε είναι άλλο θέμα όσον αφορά το συμβιβασμό. Αν υπερψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε είναι άλλο θέμα. Αλλά με μια προφορική τροποποίηση, αν κάποιο είναι εναντίον, τότε δεν μπορεί να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση. Αυτό λένε οι κανονισμοί. Το κατάλαβα. Χωρίς την προφορική, γιατί αντιτίθεστε στην προφορική. Εντάξει, έτσι το κατάλαβα, λέει η Πρόεδρος. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Je Ψηφίζουμε. Επί της 13 το R τεσσάρων πολιτικών ομάδων χωρίς την προφορική υπέρ. Υπέρ της R, της, του συμβασμού, κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Tout le monde a pu voter Μπόρεσαν να ψηφίσουν όλοι, λειτουργούν όλα τα μηχανήματα. Πέρες ψηφοφορία 24 υπέρ 22 κατά εγκρινέται με την ίδια πλειοψηφία. Φτάνουμε λοιπόν μετά την παραγραφό 13 στην παραγραφό 19 της Επιτροπής ΦΑΜ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 308 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να το επαληθεύσουμε γιατί δεν ψήφισαν όλοι. Άρχεται η ψηφοφορία για την 308. Tout le monde a pu voter le vote est clos. 24 22 υπέρ, 22 κατά, η ίδια γνωστή πλειοψηφία περνάει τις ιδέες της. 38 ε, εγκρίνεται, 309 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 συμβεβαστική S από τέσσερις ομάδες με προφορική τρόπο τροπολογία ή δεν υπάρχει αντίθεση σε αυτή την τροπολογία. Ψηφίζεται λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε με στην 3.15 της κυρίας Τσίμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.16 του συγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.17 κυρία Άρκιν και άλλοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.18 κυρία Πλάμ υπέρ 8, κατά αποχές εγκρίνεται 3.19 κυρία Μβαρόιτεν και λοιποί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 παραγραφός 15 συμβιβαστική υπέρ α, 3.21 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 322 του κυρίου Έλμερ υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβιβαστική τε από πέντε ομάδες με προφορική τροπολογία δεν υπάρχει αντίθεση προς την τροπολογία ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 333 της κυρία Δελή. Ψηφίζουμε το πρώτο κομμάτι του κειμένου, την αρχή του κειμένου, έως το threatened with eviction. Υπέρ αυτού του προτιμήματος κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο κομμάτι υπέρ κατά οι αποχές απορρίπτεται 3, 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3, 36 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.37 της κυρίας Καρυμαντέλη υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Για την 3.37 άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας, 24 υπέρ, 22 κατά, πάντα τους ίδιους αριθμούς έχουμε. 3.38 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται 339. Παράγραφος 16 για διαγραφή 339 και 340 υπέρ. Κατά υποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική U από 5 ομάδες με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.47 της κυρίας Ντέλη και Λαμπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.48 του κυρίου Κώσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17 συμβιβαστική Β από 5 ομάδες με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 7 της Επιτροπής ε, Κουλτούρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 της ίδιας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 355 του κ. Νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο εισηγητής είναι υπέρ των όλων των υπολοιπών τροπολογιών αυτής της παραγράφου. Δεν μπορούμε να τις ε, ψηφίσουμε μαζικά. Όχι, δεν ε, συμφωνούν όλοι. 356 της κ. Νταρντέν υπέρ, κατά, αποχές. Θα υπαλληθεύσουμε για 356. Le vote est ouvert. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. 25 υπέρ 20 κατά εγκρίνεται 357 του κυρίου γιαρικη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 358 του κυρίου Φουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 260 ροντζουλί υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 262 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 261 της κυρίας Ντέλη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 359 Φιγκερέδο και άλλων υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 363 πλάμπ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 364 χάρκιν και άλλων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 365 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18, 367 πιτσότο υπέρ, κατά απο, αποχές απορρίπτεται. 367 Χέλμερ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. W, Συμβιβασμό τεσσάρων πολιτικών ομάδων με μία προφορική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εξ, τροπολογία συμβασμού τεσσάρων ομάδων με προφορική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα, όλος ευνηδίως η 264 καταπίπτει. Άρα 377 καρυμαντέλη υπέρ. Κατά. Αποχές θα επαληθεύσουμε. 379. Επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφιζα όλοι. Πέρασε. 19 pour 26. 19 υπέρ 26 κατά. 380 χάρκιν και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 381 εισηγητή, του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Μία τροπολογία 382 υπέρ, κατά. Α, καταπίπτει, με συγχωρείτε. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό ε, Y τεσσάρων ομάδων με προφορική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα φτάνουμε μετά την παράγραφο 19, 390 κόζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 391 λίν υπέρ κατά δεν ψηφίζεται πια. 391 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 393 ροντζούλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνετε 394 κόζα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 495 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 496 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράφρος 13 γυναίκες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στα έχοντας υπόψη μετά το 2, 3 τροπολογίες, 1, 2, 3 παρόμοιες. Ε, τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 5 της κυρίας Λίν υπέρ. Όχι. Κατά. Θέλετε να ψηφίσετε για την 5. 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι Ιωβίνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει μία χωρίς αρρύθμιση. Κύριε Ορή, σας ακούω. Από ό,τι μπορώ να δω, ε, η ένα, δύο, 3, α, μόνο το, οι 2 και 3 είναι ταυτόσιμες και το 1 είναι διαφορετικό. Αλλά εδώ λέει 1 και 3 ότι είναι ταυτόσιμες, identical. Εάν δεν είναι όλες ταυτόσιμες, θα ήθελα να ψηφίσουμε ξεχωριστά και πρώτα την 1. <laughs> le vie istruttrice delle cose di merito da Mobi. The reason, Madam, is that Mr. Jovan and myself. Ο κύριος Γιώβεν και η ίδια ο λόγος τον οποίο έχασα την αρρύθμιση είναι η τροπολογία 6, αλλά ο κύριος Γιώβεντα και εγώ υποβάλαμε την τροπολογία μαζί και γι' αυτό είναι στη λανθασμένη θέση. Ωραία. Να τα δούμε ένα-ένα. Υπάρχουν διαφορές στη σύνταξη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 1, 2 και 3, γιατί η μόνη διαφορά που βλέπω το ντρουά, το δίκαιο, είναι με κεφαλαίο ή με μικρό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό απαιτεί ξεχωριστή ψηφοφορία. Αν το θέλετε όμως θα γίνει. Δεν είναι επαρκή σε διαφορά. Αν υπάρχουν άλλες διαφορές θα ήθελα να με διαφωτίσετε. Εσείς που το γνωρίζετε και αν το γνωρίζετε. Okay. επειδή η γαλλική έκδοση είναι πιο καλή και επειδή όλοι οι συντάκτες είναι γαλλόφωνοι, το θέμα έχει λήξει. Επί της ε, τροπολογίας Harkin, εδώ υπάρχει ένα λάθος παρουσίαση στον κατάλογο ψηφοφοριών και άρα οι συντάκτες είναι Γιώβιν και Χάρκιν. Έτσι δεν είναι κυρία Χάρκιν. Άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Ορί, ο κύριος Ορί. Bien. Alors, nous en venons... Δεν έχει να πει τίποτα. Ωραία. Μετά την αιτιολογική σκέψη 4, 7 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 8 του εισηγητή, που θα πρέπει να μπει αλλού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 του κυρίου Χέλμερ που θέλει τη διαγραφή της αιτιολογικής σκέψη 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την 9 τροπολογία 10 και 11 που είναι παρόμοιες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Μετά το 12, 12 της κυρίας Κιγκαγκένς υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το 16, 13 του εισηγητού και άλλων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη 18, τροπολογία 14, Καρή Μαντέλη και άλλων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24, προφορική του εισηγητή, όπου γίνεται μία προσθήκη σε ένα, για ένα ψήφισμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15. Καρίμα Ντέλ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη 25, 16 ε, Ντέλη και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 κίνγκα, με συγχωρείτε, 17 υπέρ κίνγκα Guns υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την ετολογική σκέψη 25, προφορική του εισηγητή, δεν αντιτίθεται κανείς, ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά άλλη μία προφορική του εισηγητού, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική μπορούμε να πάρουμε όλη την αιτιολογική της Επιτροπής ΦΑΜ. Τέσσερα 6, 7, 8, 9 και 11 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εκτιμώντας α, συμβαστική ζ, 5 ομάδων με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά συμβιβαστική α δεν γνωρίζω τους συντάκτες, τροπολογία προφορική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στο εκ, την, ε, τροπολογία 30 που καταπίπτει. Περνάμε στο εκτιμώντας β. Συμβιβαστική ΒΒ. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά από τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική σε, σε στην, από πέντε ομάδες με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την ιδεολογική σε τροπολογία 47 από καταπίπτει, 48 της κυρίας Τσίμερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 51 του κυρίου Έλμερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 52 Φιγκερέντο υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε για την 52 τροπολογία της αιτιολογικής σκέψης σε B άρχεται κλείνει ψηφοφορία 23 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται Εκτιμώντα D, τροπολογία 53 πίπτη, συμβιβαστική D, 5 ομάδων με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην 58 τροπολογία των κυρίων Μπεναμίας και λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 της κυρία Λόπε Φωντανιέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 της κυρία Τσίμερ υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε για, το, για την τροπολογία 63 ψήφισαν όλοι Κλείνει η ψηφοφορία. 18 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Θέτουμε σε ψήφο λοιπόν την προπολογία 65 της κυρίας Τσίμερ υπέρ. 64 ε, συζητώ συγγνώμη. Ε, συγγνώμη, η 65 της κυρίας Τσίμερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Την 65 μπορεί να ψηφίσουν όλοι για την τροπολογία 65, κλείνει η ψηφοφορία, 18 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Εκτιμώντας ε τροπολογία 66 της κυρίας Μπιτζότο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, συμβιβαστική ε ε 5 ομάδων με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69 της κυρίας Ρενιέρ και λοιπόν υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε την τροπολογία 69. Ψήφισαν όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. 17 υπέρ 27 κατά απορρίπτεται σαφώς 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας F71 της κυρίας Μπιτζότου για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική FF πέντε ομάδων με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στην 78 της κυρίας Μπιτζότο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική GG με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 84 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική HH 5 ομάδων με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας H τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 γιωταγιωτα πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 94 του κ. Έλμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 96 του κ. Νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική JJ ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 95 λοιπόν καταπίπτει 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 του κ. Μπουλόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 του ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία συνδυασμού διπλό κάπα πέντε πολιτικών ομάδων με μια προφορική υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 105 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κάπα 106 του κυρίου Χέλμερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβασμού διπλό L, πέντε ομάδων με μία προφορική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα τώρα φτάνουμε εσίως σε τρία έχοντας υπόψη της ΦΑΜ να τα δούμε unblock. DF και υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 113 Helmer υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114 στο Ελ Λόπε Φοντέν και άλλων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 Μπεναμίας και άλλων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. M, διπλό M, 5 πολιτικών ομάδων με προφορική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 123 της κυρίας Μπιτζότο, διαγραφής υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Διπλό N, συμβιβασμός 5 πολιτικών ομάδων με προφορική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το 1.128. 128 Λεϊαρίκ και άλλων, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο όμικρον 129 της κυρίας Μπιτζότο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Π, 130 Μπιτζότο, για διαγραφή υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβασμός διπλό ομίκρον πέντε πολιτικών ομάδων με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Μετά το P133 της κυρίας Ντέλη και άλλων υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουν. Επαληθεύουμε την 133. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τι Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 23 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται με μία πλειοψηφική 134 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 Χάρκιν και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το π 137 του εισηγητή και άλλων υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε. 137 ψηφίζουν. Tout le monde le vote est clos. 23 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται. Και τώρα φτάνουμε ε, στην ηλεκτρονική επαλήθευση του σχεδίου. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εσίως, οι 34 υπέρ, 5 κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Alors, nous en venons au point 13 de notre... Σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Και θα ψηφίσουμε... Μια σειρά τροπολογιών που θα υποβάλουμε ως αμπλουά στην ΑΦΕΤ σε σχέση με την αίτηση της Κροατίας για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Παράγραφος 1. Πριν από την παράγραφο 1, ησυχία παρακαλώ, τροπολογία 1, τέλη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2, συμβιβασμός α δύο πολιτικών ομάδων με μία προφορική. Δεν αντιτίθεται κανείς στην ε, προφορική. Α, συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Συμβιβασμός Α. Δύο πολιτικών ομάδων. Άρα καταπίπτει η προφορική. Συμβιβασμός Α. Υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 2, τροπολογία προφορική της κυρίας Γιασλοβιέτσκα. Αντιτίθεται κανείς στην προφορική. Όχι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, τροπολογία 3, θέρκας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, συνδυασμός β. 5, δύο ομάδων ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το παράγραφο 5, τροπολογία 5. Σέρκα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Κορνέλισεν υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. 6. Της κυρίας Κορνέλισεν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Tout le monde a pu voter Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 21 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο... Η κυρία Τσίμερ. Αν θέλω την προφορική τροποποίηση να πω ότι διαφωνώ με αυτήν. Δεν συμφωνώ να τεθεί σε ψηφοφόρια. Καταπίπτει λοιπόν. Δεν έχουμε τελική ψηφοφορία 16 τροπολογίες θα υποβληθούν εξ ονόματός μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια έχουμε μία τελευταία ψηφοφορία που αφορά την επιστολή σε σχέση με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με βάση μια αίτηση της Γαλλίας που υπέβαλε η Γαλλία για την επιχείρηση Ρενό Υπάρχει τροπολογία συμβιβασμού των σοσιαλιστών και του ΕΛΚ σε σχέση με την οποία θα ήθελα να σας υποβάλω μία προφορική τροπολογία διότι λείπει ένα άρθρο. Και η τροπολογία είναι ζητά την Επιτροπή Προπολογισμών να αναστείλει στείλει να βάλει κατά μέρο ένα ε, χρηματικό ποσό μέχρι ότου γίνει ε, έλεγχος των λογιστικών από την Κομισιόν. Νομίζω κανείς δεν αντιτίθεται. Όχι, όχι. Δεν συμφωνούμε, λέει ένας ομιλητής. Κύριε Καμόρ, νομίζω ότι δεν ε, καταλάβατε ότι κάνω χιούμορ, διότι η τροπολογία συμβιβασμού όπως έχει συνταχθεί έχει ένα λάθος, Έχει ένα λάθος, λείπει ένα άρθρο που είναι η μνήα του A και κλπ. Δηλαδή θα προσθέσουμε μόνο το α. Ας, συντάξουμε καλά λοιπόν το κείμενο στην αγγλική και ας μην την κατέχουμε καλά. Άρα δεν γίνεται δεκτή η ε, αίτησή σας. Εν πάση προτείνω να ψηφίσουμε επί της επιστολής με αυτή την τροπολογία συμβιβασμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας γίνει επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία, αρχίζει η ηλεκτρονική. Tout le monde a pu voter? Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται η επιστολή με 38 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά και μία αποχή. Ωραία, τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ και όπως συμφωνήθηκε χτες θα περάσουμε στο θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης και σας παρακαλώ ησυχία και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κρίστεσεν, ο οποίος θα μπορέσει να λάβει το λόγο στα δανέζικα για το ενωσιακό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Έχετε το λόγο και μπορείτε να μιλήσετε στη μητρική. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι μία έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Η η οποία πήγε στην Επιτροπή Νομικών ε, Υποθέσεων είναι γνωμοδότησή μας εις απάντηση της Πράσινης Βίβλου για την ε, εταιρική διακυβέρνηση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε υπερβολικά δικητικό διοικητικό ε, βάρος ε, στην εταιρική διακυβέρνηση. Τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικοί έχουν μία ευθύνη ε, στην εταιρική διακυβέρνηση, αλλά επίσης πρέπει να λάβουν υπόψη και την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά το βασικό είναι η ευθύνη των εργοδοτών προς την ευημερία των εργαζομένων και η έλλειψη ευθύνης και η ανάληψη ευθύνης ήταν, είναι μία, ένα από τα αίτια της σημερινής δινής κατάστασης. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μια ενα απο τα αιτια της σημερινή δινης καταστασης διακυβέρνηση ε, σε μια εταιρεία δεδομένου ότι η επένδυση στο εργατικό προσωπικό είναι μακροπρόθεσμη η διοίκηση ε, είχε μία στενόμυαλη ε, προοπτική ε, κέρδους μέχρι τώρα, επικεντρωνόταν υπερβολικά στο κέρδος, ενώ αυτή τη στιγμή θέλουμε να εφαρμοστεί μία ολοκληρωμένη εταιρική διακυβέρνηση, η οποία να λαμβάνει υπόψη και κοινωνικές και ηθικές αξίες. Δεν είναι δυνατόν να στοχεύουν μόνο στο βαχυπρόθεσμο κέρδος οι διοικήσεις των εταιριών. Η διοίκηση θα πρέπει να εστιάζεται στην ε, αηφόρο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ε, και ευημερία της εταιρεία και να εκτελεί υπεύθυνε και ησικές επενδύσεις αντί να επικεντρώνεται σε και κερδοσκοπικές ενέργειες. Οχτώ σημεία αναφέρονται στην έκθεση 8 προτάσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια, στη σταθερότητα της του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και στις κοινωνικές και ηθικές αξίες. Η εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεων με τους εργαζομένους, και ε, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι συμβάλλουν και εξαρτώνται ιδιαίτερα από την επιτυχία και την απόδοση της εταιρεία. Και η Κομισιόν αυτό δεν το αναφέρει καθόλου στην πράσινη βίβλο, διότι οι εργαζόμενοι μπορούν να παίξουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη των εταιριών. Επίσης θα πρέπει να επιτρέπουμε τη συμμετοχή και να σαρίνουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε αυτό θα πρέπει να είναι μια υποχρεωτική ε, κατευθυντήρια γραμμή και να το ασπαστεί η διοίκηση των επιχειρήσεων δεδομένου ότι μόνο όφελος μπορεί να αποφέρει συμμετοχή εργαζομένων με διαφορετικές δεξιότητες ε, στη ε, διοίκηση της εταιρείας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, επίσης, ε, θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη να μην υπάρχουν προσκόμματα όσον αφορά το πακέτο ε, των αμοιβών. Αυτό το θέσαμε υπόψη ε, και στις, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ότι πρέπει να δίδονται ευκαιρίες απόκτησης μετοχών της εταιρεία σε ένα ποσοστό μέχρι 50% η διανομή των μετοχών, των μετοχών μεταξύ των εργαζομένων πιστεύω ότι είναι μια θετική ιδέα, μια, μια θετική ε, πράξη, ε, διότι ε, αυξάνει τα κίνητα εργασίας και μειώνει τους κινδύνους και γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται κάθε τριετία μια αξιολόγηση των εισαγμένων εταιριών και αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές Κομισιόν στην Πράσινη Βίβλο. Πέραν αυτών όλα τα μέλη ε, το, του, της διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να δημοσιεύουν τα επιχειρησιακά τους, ε, τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες που εμπλέκονται, τι ενδιαφέροντα έχουν και τι θέσεις έχουν. Ε, έτσι ώστε πιστεύω ότι θα έχουμε μια επικοδομητική, θα γίνει επικοδομητική δουλειά σε αυτό το θέμα και θα συνεργαστώ ε, πολύ καλά με τους Κιώδης, η κυρία Μπάουερ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Δεν ήταν καθόλου εύκολη η δουλειά του διότι η βίβλος για την ε, εταιρική διακυβέρνηση και σε σχέση με την ε, ανάγνωση το κείμενο δεν είναι καθόλου ευανάγνω, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και η ε, εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι ο κύριος πυρήνας αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Ωστόσο όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα σημαντικό στοιχείο σε σχέση με τις τροπολογίες που κατατίθενται σε αυτή τη γνωμοδότηση σε αυτήν την έκθεση. Πρώτα απ' όλα το θέμα των αμοιβών. Μεγαλύτερη διαφάνεια χρειάζεται, πρέπει να πω. Και οι αμοιβέ θα πρέπει να συνδέονται πιο στενά και να βρίσκονται σε αναλογία με την κερδοφορία της ε, εταιρεία. Δεύτερη παρατήρηση, η συμμετοχή γυναικών. Η συμμετοχή των γυναικών σε τέτοιου είδους ε, εταιρικά συμβούλια. Η Επίτροπος Ρέντινγκ, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και σαφή πρωτοβουλία ανέλαβε επί του θέματος αυτού. Και τρίτον, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις προτάσεις ε, του εισηγητού επί του ότι η πράσινη βίβλος δεν τονίζει επαρκώς, καθόλου δεν τονίζει το θέμα του κοινωνικού διαλόγου και συναφών θεμάτων. Και αυτό είναι κάτι που δίκαια υπέστη επικρίσεις από πλευράς εισηγητού. Ευχαριστώ. Κοφεράτη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο για την πρότασή του. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε έναντι της Κομισιόν. Ε, δηλαδή, από πλευράς επιχειρήσεων, να ζητήσουμε να υπάρχει διαφάνεια. Να έχουμε όλο το φάσμα στοιχείων που προβλέπονται. Εάν κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση θα επιλύσουμε και το θέμα της διαφάνειας και το θέμα αντιμετώπισης ε, όλων των stakeholders. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε την επιχείρηση και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Θα πρέπει να υπάρχουν συμμετοχικές διαδικασίες οι οποίες ε, προέρχονται από το ε, σχέδιο αμοιβών, από το σχήμα αμοιβών. Δεν καταλαβαίνω γιατί λοιπόν ένας εργαζόμενος που διατρέχει τον ε, κίνδυνο να αλλάξουν οι σχέσεις του Άρδιν με την επιχείρηση. Δηλαδή, αν κλείσει η επιχείρηση, δεν θα έχει ούτε εργασία, ούτε αμοιβή. Και άρα υπάρχει και ένας ε, επόμενος, ε, επόμενο βήμα, δηλαδή σε περίπτωση πτώχευσης αυτής της επιχείρησης ο εργαζόμενος θα υποστεί διπλό, διπλή ζημία σε σχέση με την εργασία του και σε σχέση και με το μισθό του ή τις αποταμιεύσεις του. Και δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να υπάρξει συμφωνία, ε, αυτή η σχέση δηλαδή μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων. Είναι σαν να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ευχαριστώ. Κάποιος ε, άλλος που θα ήθελε να μιλήσει. Ναι, παρακαλώ. Philippe de I'm εισηγητής από πλευρά της ομάδας μας θέλω να ευχαριστήσω και εγώ Κρίστενσεν για αυτή την έκθεση και τη δουλειά που έχει επενδύσει. Μπορείτε όμως να φανταστείτε, δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλα τα σημεία που προνοιτερική διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι θέμα της ίδιας της εταιρείας. Εδώ ε, το, η κύρια πρόταση είναι από πλευρά μου ότι εγώ δεν είμαι υπέρ του να δεσμεύεται η νομοθεσία ως προς αυτό. Είμαι περισσότερο υπέρ ενός διοντολογικού κώδικα που θα πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις και θα είναι προς όφελος των επιχειρήσεων να ακολουθούν αυτόν τον διοντολογικό κώδικα από πλευρά τους. Πρώτη μου παρατήρηση αυτή. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν μπορούμε ισοπεδωτικά να υιοθετούμε μια ε, πρόταση ότι μία και ε, ενιαία πρόταση θα πρέπει όλων των εταιριών να εφαρμόζεται. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, ε, πολυεθνικές, υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν ισοπεδωτικά να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά όσον αφορά τους εμπλεκόμενους και τους εργαζόμενους να υπάρχει ένα στενό κορσές υποχρεώσεων που θα είναι ίδιος για όλες τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να είμαστε πιο ελαστικοί, πιο ευέλικτοι στην προσέγγιση μας για κάθε είδου εταιρεία ξεχωριστά ανάλογα με τις διομορφίες της και λαμβάνοντας υπόψη και τις μελλοντικές ανάγκες αυτών των εταιριών. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να προτείνω μια μη δεσμευτική, εθελοντική, εθελούσια βάση για ένα διοντολογικό κώδικα για τις ε, εταιρείε όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και έτσι να λειτουργήσει αυτό από πλευρά ε, των κρατών. Δεύτερον, όσον αφορά την πολιτική για αμοιβέ, όπου ο εισηγητής προτείνει απαγόρευση όσον αφορά τις ε, μετοχές και τις ε, δυνατότητες ε, απόκτησης μετοχών. Θα έπρεπε οι εταιρείε να μπορούν σε σχέση με την αντίστοιχη επιτροπή να ε, διαμορφώνουν το τι, μπορεί, τι θα μπορεί να γίνεται και τι θα, ποιες δυνατότητες θα είναι ανοιχτές για την πολιτική αμοιβών από πλευρά της εταιρείας. Και όσον αφορά και τις εισηγμένες εταιρείε, αλλά αυτό πάλι δεν θα πρέπει να επιβαρύνει ε, ή να ε, είναι ε, περιοριστικό για μικρές εταιρείε. Συμφωνώ με άλλα σημεία για τη σημασία που έχει η διαφάνεια όσον αφορά την, και την πολιτική διαμόρφωση και αντιμετώπιση κινδύνων και όσον αφορά και τα μέλη του Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου και την σημασία, τη σπουδαιότητα του να επεξηγούνται αυτά τα πράγματα. Επιμέρους κάποια επιπρόσθετα στοιχεία που θεωρώ ότι μπορεί να είναι ενδιαφέροντα από πλευρά μου. Η ισοπεδωτική εφαρμογή μια αρχή εφόλων των επιχειρήσεων δεν νομίζω ότι είναι σωστή προσέγγιση. Θα πρέπει να δούμε τις υφιστάμενες συστάσεις ε, για την εταιρική διακυβέρνηση που ήδη υπάρχουν και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Και εδώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών, διαφορών στις πρακτικές ε, που υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών εταιριών όσον αφορά τα κρατη και στα διοικητικά συμβούλια και στην εκπροσώπηση και συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά τα συμβούλια. Υπάρχουν τελείως διαφορετικές δομές ε, και εκπροσώπηση ανάλογα με τις χώρες μας και δεν θα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα ε, που αναφύονται με μία ισοπεδωτική προσέγγιση που θα εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείε. Πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι, πιο ε, ε, ελαστικοί. Προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία με τον εισηγητή να, βρούμε τους, να βρούμε τους καλύτερους συμβιβασμούς. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κύριε Ντεμπάκερ. Υπάρχουν άλλε αιτήσει ομιλία. Δεν βλέπω να σημαίνει κάτι τέτοιο. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους προλαλήσαντες για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους, τα οποία σίγουρα είναι πολύ χρήσιμα και ε, θα τα μελετήσω για την κοινή πρόταση που θα υποβληθεί. Ε, το θέμα της πολιτικής των ε, μισθών και αμοιβών πρέπει να είναι διαφανές και ανοιχτό προσβάσιμο σε όλους από την Αλδε τώρα τα σχόλια ε, και τις αντιρρήσεις ε, για την ε, μείωση του, του δικαιώματος αγοράς μετοχών, δικαιώματος αγοράς μετοχών. Εδώ μιλάμε για την προσφορά μετοχών σε, σε τράπεζες οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί ή βούλιαξαν λόγω των κινδύνων που ανέλαβαν. Την τελευταία φορά μόνο τρεις καταψήφισαν την απαγόρευση της δυνατότητας δικαιώματος αγοράς μετοχών. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να απαγορευτεί, εγώ λέω ότι θα πρέπει να ελεγχιστοποιηθεί η δυνατότητα δικαιώματος αγορών μετοχών και ιδανικά να, καταργη, να καταργηθεί σταδιακά δεν μπορούμε να καταργήσουμε τους ε, κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι έως 50% μπορούν οι εργαζόμενοι αντί αμοιβή να αγοράσουν, να λάβουν δικαιώματα μετοχών. Ε, ανάλογα βεβαίως με την αξιολόγηση της απόδοσης τους. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Μπάουερ για τις ε, γυναίκες και τη συμμετοχή τους. Μου είπε η γραμματεία ότι Οι ποσοστώσεις δεν είναι δική μας αρμοδιότητα στην Επιτροπή Απασχόλησης. Γι' αυτό πάντοτε αναφέρομαι στην ε, ε, διάκριση του φύλου, στην ε, συμμετοχή και των δύο φύλων, εννοώντας βεβαίως και την συμμετοχή των γυναικών. Για τον κοινωνικό διάλογο Συμφωνώ ότι αυτό λείπει προς το παρόν από την έξι τη Κομισιόν, αλλά και χρειάζεται να προσθέσουμε μερικέ πτυχέ ε, για τον κοινωνικό διάλογο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αυξάνει την κοινωνική ευθύνη των εταιριών. Ο κύριος Κοφεράτη, ο καλός μου συνάδελφος, δεν ε, είναι υπέρ ε, των μετοχών ή των εθελοντικών, της εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο. Εδώ έχουμε μία διαφοροποίηση της κατάστασης σε κράτη-μέλη. Ε, στη, στη δικιά μου χώρα και στις εταιρείε που ξέρω, πάρα πολλοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν αυτή την οψιόν, αυτή τη δυνατότητα να πάρουν μετοχές, διότι διότι πιστεύουν ότι αποτελεί και ένα κίνητρο βελτίωσης και της εταιρείας και των, ε, της εργασίας τους. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι θετικό, μια θετική ιδέα. Δεν πιστεύω ότι οι μετοχές πρέπει να αντικαταστήσουν ένα τμήμα των μισθών και αμοιβών, έτσι ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθούν οι αμοιβέ του προσωπικού, ε, διότι τι θα γίνει όταν η εταιρεία χρεοκοπήσει. Όμως πιστεύω ότι είναι μια ένας καλός, ένας σωστός τρόπος ε, συμμετοχής των εργαζομένων. Συμφωνώ ότι, δεν θα, ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα και με το μέγεθος των εταιριών. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις σε μικρές και μεγαλυ, ή μεγαλύτερες εταιρείε, διότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε υπερβολικά μικρότερες εταιρείε με αυτή τη διαδικασία. Ε, όταν ο συνάδελφος από την ΑΛΔΕ λέει ότι δεν θέλουμε οι κανονισμοί αυτοί να είναι υποχρεωτικοί, γιατί καλύτερα είναι να έχουμε έναν κώδικα δεοντολογίας, μα και αυτός θα είναι δεσμευτικός, δεν θα είναι. Πώς λοιπόν, ε, τι συμβαίνει λοιπόν στις εταιρείες οικονομικού περιεχομένου που λειτουργούν σε παγκόσμιο περιβάλλον. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζονται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο υποχρεωτικό χωρίς ε, να αυξηθεί υπερβολικά το διοικητικό άχθος. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. και για την γνωμοδότησή σας. Βάσει αυτών δίνουμε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, δυστυχώς μικρή όπως ε, πολύ συχνά, μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, 12 η ώρα. θα τις εξετάσουμε 7 ή 22 Νοεμβρίου για να τις ψηφίσουμε στις 5 Δεκεμβρίου. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο τη σημερινή διάταξη και όπω συμφωνήθηκε χθε θα περάσουμε στο σημείο 16. Έτσι δίνω λοιπόν ε, το λόγο στο συναδελφό μα ε, Σβέν Γκόλντ όσον αφορά το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα, ήδη είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Εξίσου ευχαριστώ επίσης και τους σκιώδεις εισηγητές των διαφορετικών κοινοβουλευτικών ομάδων. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση, υπήρξε εκεί μια ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ την Άντια Χίρσα από τους φιλελεύθερους και από πλευρά τη ε, δουλειά που είχε γίνει από τη Σοφή. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Εδώ ουσιαστικά είχαμε μια παράλογη κατάσταση. Εργαζόμαστε για μια μεταρρύθμιση που για ένα ε, ταμείο το οποίο δεν ε, ε, έτυχε κάποιας υποστήριξης ή προαγωγής που είναι όμως η μόνη μορφή οικονομία από πλευράς οικονομίας και κοινωνικής οικονομίας να δραστηριοποιούνται τα, οι συνεταιρισμοί Πολλοί συνάδελφοι σε γραπτές επεξηγήσεις εξέφρασαν παράπονα ότι εξακολουθούν για ενώσεις, συλλόγους και αμοιβέ τέτοιες ενώσεις, συνεταιρισμούς δηλαδή, δεν να μην υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο ευρωπαϊκά. Και είναι προφανές πλέον ότι ο τομέας των συνεταιρισμών και της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας συνολικά παρέχει ένα μεγάλο δυναμικό για την οικονομία και μεγάλη δυνατότητα δραστηριοποίησης. Ε, έτσι ακολουθούνται ταυτόχρονα διτοί στόχοι, ένας διπλός στόχος. Αφενός ε, να μπορέσουν να παρέμβουν ε, όσο το περισσότερο στην αγορά και οικονομικά και να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν τους εργαζόμενους, τα μέλη τους. Και αυτή, αυτός ο διπλός στόχος είναι ακριβώς που οδήγησε στο ότι πάντα να υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη, ευρύτατη υποστήριξη για αυτούς τους στόχους. Επανειλημμένα και στην έκθεση τα παριθμό αυτά, το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν μέτρα και πρωτοβουλίες στον τομέα των συνεταιρισμών, των οικονομικών δραστηριοτήτων, σε ενώσεις, συλλόγους και σε πολλούς άλλους τομείς τομεακά αυτής της οικονομίας, δηλαδή της κοινωνικής αλληλεγγύης, να υπάρξει υποστήριξη. Δεν θέλω να επισέλθω τώρα στα διάφορα σημεία και προβλήματα. Αν προβλήματα συμμετοχής των εργαζομένων θα πρέπει να περιορίζονται, θέλω να διευρύνουμε το θέμα στο φάσμα του πόσο το δυναμικό απασχόλησης ε, και οικονομικό δυναμικό σε αυτό τον τομέα μπορεί να ενισχυθεί, να ενδυναμωθεί. Ουσιαστικά η έκθεση έχει δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα παρουσιάζει το πρόβλημα σε σχέση με αυτή τη νομική δομή και επισημαίνει ότι αλλαγές όσον αφορά την συνδιαχείριση ή συναπόφαση των εργαζομένων είναι αναγκαία υπόθεση να διασφαλιστεί αυτή η συνιστόσα. Όμως ταυτόχρονα ουσιαστικά το αποφασιστικό, αποφασιστική σημασία πρόβλημα για την χρήση αυτών βρίσκεται στο ίδιο το καταστατικό και ζητείται να εξεταστούν τα ζητήματα και προβλήματα που υπάρχουν και αναφύονται σε σχέση με, με το καταστατικό και αυτά να επιληθούν. Και δυστυχώς είναι τόσο περίπλοκο το καταστατικό που δεν μπορεί ο τομέας να το χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά κλασική περίπτωση υπερβολικής γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Οι πραγματικά εμπλεκόμενοι στην αλληλεγγύη, δηλαδή στην κοινωνική οικονομία, δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν σωστά. Υπάρχει ο φόβος η σημερινή αυτή δομή να χρησιμοποιείται ώστε να υπονομεύονται και να περιορίζονται δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτή η νομική μορφή ουσιαστικά όμως δεν χρησιμοποιείται καν Γνωρίζουμε ότι και με άλλου είδους τέτοιες νομικές δομές υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να τα αποφεύγουμε. Εδώ ο κύριος ε, στόχος είναι να είναι θελκτικό, ελκυστικό το πλαίσιο αυτού του νομικού πλαισίου και έτσι να διασφαλίζονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων με τις ιδιομορφίες και όπως παρουσιάζονται και διαμορφώνονται στους συνεταιρισμούς. Και γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά οι εργαζόμενοι είναι συνειδιοκτήτες πολλές φορές και τίθενται ζητήματα της συμμετοχής των εργαζομένων υπό διαφορετικό πρίσμα. Αλλά εξακολουθούν αυτά τα θέματα να είναι σημαντικά. Και μετά αναφέρονται στο άλλο τμήμα οι πολλές ελλείψεις και τα προβλήματα που έχουν οι συνεταιρισμοί στην Ευρώπη που είτε την χάνουν αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης, δυσμενώς δηλαδή αντιμετωπίζονται, είτε δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη για αυτού του είδους ε, δράσης. Και γι' αυτό πιστεύω είναι σημαντικό εμείς, ε, όπως και στο σύνολο της έκθεσης, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια ευρεία πλειοψηφία, να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν, να εφαρμόσουν τα διαφορετικά αυτά μέτρα, ώστε να υπάρξει ενδυνάμωση της κατοχήρωσης, ε, της ε, ε, συμμετοχής της κοινωνικής αλληλεγγύης λαμβάνοντα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες, οι όροι και προϋποθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρονται έτσι νομικά και να διασφαλίζονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχω υπόψη σε συνεργασία με τους ε, σκιώδεις συζητητές να προχωρήσουμε θετικά μέσα σε ένα επικοδομητικό πλαίσιο στη συνεργασία μας και όχι μόνο να έχουμε μια ωραία έκθεση ιδείας πρωτοβουλία, αλλά στη συνέχεια να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα παρακολουθώντας το και συνοδευτικά βλέποντας πώς μπορούν να ενδυναμωθούν όλα αυτά. Και από πλευράς του κυρίου Μπαρνιέ θα ήταν ευκταίο με τις δράσεις του που, έχει, έχουν ένα πιο ε, θετικό και επιθετικό χαρακτήρα αλλά και η υπόλοιπη Επιτροπή να εμείνει ώστε ε, τα δικαιώματα αυτά των εργαζομένων μέσω των διαφορετικών γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των διαφορετικών τομέων να προαχθούν. Αυτό είναι ένας από τους λόγους, επειδή δεν έγινε αυτό, το ότι δεν έχουν προαθεί αυτά. Και περαιτέρω προτάσεις που πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε σχέση με τα 12 σημεία από το 2004 για τους συνεταιρισμούς μόνο εν μέρη εφαρμόστηκαν, μερικώς και θα πρέπει ως Κοινοβούλιο να εμείνουμε και να επιμείνουμε να πιέσουμε ώστε να υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά αυτό είναι προς το συμφέρον της απασχόλησης και προς το συμφέρον της δημοκρατίας ήδη στην οικονομία ευρύτερα. Και νομίζω ότι έτσι έχουμε μια καλή ομάδα ώστε με ευρεία πλειοψηφία και συνενετικά να προχωρήσουμε. Προσβλέπω στις παρατηρήσεις σας και είμαι βέβαια ότι υπό το πρίσμα του συμβιβαστικών προσπαθειών θα βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Ρέινερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, όχι για την παρουσίαση μόνο της έκθεσης, αλλά και για τον τρόπο όπως μέχρι σήμερα αναπτύχθηκε η συνεργασία και εξελίχθηκε η συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό, το ότι είχαμε την ευκαιρία ήδη πιο πριν προηγούμενα να συλλέξουμε και να ανταλλάξουμε ιδέες και να συζητήσουμε για πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται. Θα ήθελα τώρα στη συνέχεια, ας το πω έτσι, να προχωρήσω πιο πέρα. Και αυτό επειδή η προσέγγιση όσον αφορά τη, τα θέματα υποσυζήτηση ήταν αρχικά εκείνη ώστε για αυτούς τους συνεταιρισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν γίνονται πολλά. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πρότυπο να θεωρηθεί ως το πιο επιτυχημένο πρότυπο στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Γι' αυτό είναι σαφές και ε, έχει νόημα και νομιμοποιούμεθα να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Εν μέρη κράτησε ε, μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά όμως και την ποιότητα αυτές τις αρχές. Ως προς αυτά θα έπρεπε κάποιες επιφυλάξεις ε, να αναφερθούν και κάποια ε, στοιχεία να τονιστούν. Πρώτα απ' όλα κάνω λόγο για τη δική μου τη χώρα, την Αυστρία φυσικά και θα ήθελα εκ προημίου να αναφέρω ότι οι διαπιστώσεις και προτάσεις κινούνται προς μια ενισχυμένη ε, δυνατότητα χρησιμοποίησης, χρήσης και εφαρμογής ε, αυτού του προτύπου ε, συνεταιριστικής δραστηριοποίησης και θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση. Πολλά μπορούν και πρέπει να γίνουν. Όμως οι συνεταιρισμοί με διαφορετικό τρόπο υποστηρίζονται και χρησιμοποιούνται αναχώρα. Έχουμε στην Αυστρία ουσιαστικά ένα μεγάλο συνεταιρισμό που δραστηριοποιείται ε, αντίστοιχα, όμως αυτό δεν γίνεται σε σχέση με την εφαρμογή ενός ε, προτύπου ε, ευρωπαϊκού, αλλά υπάρχουν για παράδειγμα υπομορφή ε, ε, μετοχικών εταιριών άλλες επιχειρήσεις ε, που δραστηριοποιούνται και οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και αν υπάρχει για την χρήση του ευρωπαϊκού προτύπου θα πρέπει να λαμβάνονται αυτές οι ιδιομορφίες υπόψη. Δεν είναι όλες, όλοι οι συνεταιρισμοί παν, πανομοιότυποι. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες δραστηριοποίησης. Και περνάω στο επόμενο σημείο. Θα έπρεπε να είναι στόχος ε, που ε, θα ήταν σκόπιμος να γίνει πιο θελκτικό αυτό το πρότυπο, το συνεστεριστικό πρότυπο. Δεν είναι όμως αυτός σκοπός αυτό, δεν μπορεί να είναι αυτός σκοπός και έτσι προχωρώ σε σχέση με τις προτάσεις για το καταστατικό. Πρέπει να προσέξουμε να απλουστευτούν αυτές, ε, να μην γίνουν μέσα σε ένα περίπλοκο σύνθετο πλαίσιο. Γιατί, για παράδειγμα, σε σχέση και με την δυνατότητα κεφαλαίου να ληφθεί η συνιστός αυτή υπόψη. Δεν θα ήθελα σε ευρωπαϊκό ε, πρότυπο να μην ληφθεί το θελκτικό αυτό στοιχείο, ελκυστικό στοιχείο υπόψη και να έχουμε ε, υποβαθμισμένες, ε, όχι μόνο σε σχέση με τις, τη συμμετοχή των εργαζομένων με μετοχές, αλλά και με την ε, ίδια την ε, ε, ενεργό οικονομική συμμετοχή τους. Για τις προτάσεις αυτές θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό το οποίο προτείνεται και πρέπει να μεριμνήσουμε να ενδυναμώσει στις δράσεις της αυτή την πτυχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης να ληφθούν υπόψη, διότι στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας υπάρχουν, ας το πω έτσι, υπάρχει η ανάγκη να έχουμε την παρουσία πραγματογνωμοσύνης και εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τα οικονομικά θέματα. Και επίσης να λάβουμε υπόψη το ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και να προσέξουμε στις προτάσεις που τώρα κατά το μάλλον ή τον στοχεύουν στη συνδιαχείριση, απόφαση των εργαζομένων, να μην υπάρξει κάποια αντίφαση ή αντίθεση σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί, να μην είναι υπερβολικά περίπλοκες ε, και να μην επιβαρύνουν γραφειοκρατικά. Αν τα καταφέρουμε αυτά, ε, τότε η έκθεση θα μπορέσει να υποστηριχθεί από εμάς. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε σε αυτά τα στοιχεία για να το καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Χίρς. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γκίνγκοντ για την συνεργασία αυτή που ξεκίνησε και χαίρομαι και για τη μελλοντική συνεργασία. Είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ιδεολογικά ή κομματικά, αλλά πρέπει ρεαλιστικά να το αντιμετωπίσουμε. Και πρόκειται για μια σημαντική μορφή ε, δραστηριοποίησης που έχει πολλά προτερήματα σε σχέση με τους συνεταιρισμούς. Για όσους συμμετέχουν και η συμμετοχική δραστηριότητα είναι σημαντική η συμμετοχή και μπορεί να πράγματι να υποστηριχθεί και η πολυμορφία, η ποικιλομορφία των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται είναι και αυτό ένα θετικό στοιχείο. Σίγουρα κρίμα είναι το ότι δεν είναι τόσο θελκτικό αυτό το πρότυπο, δεν ήταν μέχρι σήμερα τόσο ελκυστικό. Πρέπει να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν να γίνει πιο ενδιαφέρουσα αυτή η δραστηριοποίηση και σε ένα πιο απλουστευμένο, πιο απλό πλαίσιο. Και εδώ να μην απολεστεί η απώλεια, δεν πρέπει να υποβαθμιστεί, αλλά πρέπει να αναβαθμιστεί αυτή η υπόθεση. Το υποστηρίζουμε έτσι απόλυτα. Και φυσικά το θέμα Δηλαδή, τη συμμετοχή των εργαζομένων είναι ένα σημαντικό θέμα. Πρέπει διαφορετικά να αντιμετωπιστεί από ό,τι σε άλλες ε, νομικές ρυθμίσεις, ε, νομοθετικές ρυθμίσεις. Πρέπει να το δούμε αυτό στη συνεργασία μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους που θα εμπλακούν και θα προαγάγουν αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρώτα θα μιλήσω γερμανικά και ε, ε, θα μιλήσω και γερμανικά, αλλά αν νομίζετε ότι ε, αυτή, αυτός ο συνεταιρισμός στον οποίο θα αναφερθώ είναι γερμανικός, θα μιλήσω και αγγλικά. Έχουν πιστεύω εφαρμοστεί ε, πάρα πολλές βασικές αρχές αυτού του πλαισίου, άρα θα πρέπει να στοχεύσουμε σε μια απλούστευση για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη δημιουργία περισσότερων συνεταιρισμών που παίζουν σημαντικό ρόλο και στην κοινωνική οικονομία. Γι' αυτό σας έλαβε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία, μια ενίσχυση του συντονισμού μέσα στο συνεταιριστικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας πρέπει να φροντίσει να προτείνει διατάξεις οι οποίες θα ενισχύσουν την απασχόληση ε, και, θα μπορέσουν, και να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία χωρίς προσκόμματα. Στη χώρα μου, στη Ρουμανία, ισχύει ακόμα ο νομοθεσία του 1962 ε, πολλοί συνεταιρισμοί έχουν τη δυνατότητα επέκτασης ή, περισσό, ή περισσότερης έρευνας ή πρωτοβουλίας αλλά λόγω της νομοθεσίας αυτής το συνεταιριστικό δίκτυο υποφέρει στη Ρουμανία ε, και σε άλλες χώρες. Ε, μία άλλη πτυχή του, της νομοθεσίας στη Ρουμανία είναι ότι έχει ε, ε, μία επίπτωση αρνητικών διακρίσεων. Μετά το 1989, όταν αναδιοργανώθηκε το συνεταιριστικό σύστημα, ή ο Ρουμανικός φορέας, ο οποίος ήταν υπεύθυνο για τις συντάξεις περίπου 200 συνεταιρισμών, δεν μπόρεσε να κάνει ε, μία σωστή καταχώρηση του, των παγίων του ενεργητικού και των περιουσιών των μελών, των συνεταιρισμών δηλαδή. Γι' αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την οδηγία 1432 του 2003 ε, και την αναθεώρηση του 2010 ε, που αναφέρεται στη Ρουμανία και λέει ότι η Ρουμανία έχει ένα ενεργό δίκτυο συνεταιρισμών ε, θα υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την ίδια πρωτοβουλία και θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστούμε που μας παρουσιάσετε την πραγματικότητα στη Ρουμανία, κύριε Τόμας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ ε, μου, έφτασαν η, η, μου έφτασε η παρέμβαση στα αγγλικά του συναδέλφου Ζόργα στα γερμανικά βεβαίως μέσω διερμηνίας. Ε, Σβέν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σου. Είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρον ε, τομέας. Εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε την, ε, ένα ευτυχές μέλλον σε κανένα, μια ευτυχή εξέλιξη. Εδώ δεν επιβάλλουμε τίποτα, διότι ξέρουμε ότι το όλο σύστημα των συνεταιρισμών έχει λειτουργήσει λίγαν ικανοποιητικά σε πολλούς τομείς και σε πολλές χώρες από απόψεως επιχείρησης πολλά μοντέλα είναι και λειτουργήσαν επιτυχημένα. Και στην Αυστρία και στο Λουξεμβούργο έχουμε σημειώσει επιτυχίες παρόλο που πολλές φορές δεν χρησιμοποιείς και αυτή, η δομή που πλαισιώνει του συνεταιρισμού. Πολλές φορές δεν χρησιμοποιείς και διότι ε, οδηγεί σε υπερβολική γραφειοκρατία και πολλές φορές δεν έγινε κατανοητή. Υπάρχουν λοιπόν πολλές πτυχία αυτού του πλαισίου τα οποία χρήζουν επεξεργασίες. Στο 14 λες ότι η Κομισιόν έχει κάνει μια κατανομή, μια ε, διασπορά των, εργασιών ε, και και αυτό πρέπει να το μελετήσουμε διότι όλα άπτονται της απασχόλησης ε, και γι' αυτό είμαστε αρμόδιοι. Θέλω επίσης να αναφέρω μια άλλη σημαντική πτυχή, οι συνεργάτες, η δυνατότητα συμμετοχής των συνεργατών. Αυτό πολλές φορές είναι μεγάλο πρόβλημα. Εγώ λέω πάντοτε αγαπητοί συνεργάτες, μία φορά μόνο είπα αγαπητοί σύντροφοι, οι σύντροφοι συνεταιριστέ και αυτά σε μια συνεταιριστική τράπεζα όπου χρησιμοποιούμε το γερμανικό όρο γενώσεων, δηλαδή σύντροφοι. Σύντροφοι συνεταιριστέ. Θα ήθελα πάρα πολύ να, μπορώ πολύ συχνότερα να αναφέρω τον όρο σύντροφο συνεταιριστή. Αντί συνάδελφο. Είναι νομίζω μια πάρα πολύ, ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας που δεν λειτουργεί ιδανικά προς το παρόν. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ε, οι συνεργάτες να μπορούν να συμμετέχουν ανάλογα με την ειδικότητα, ανάλογα με τις ικανότητες. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Μία άλλη πρόταση πιστεύω που κάνεις είναι πάρα πολύ σωστή. Είναι αυτό το παρατηρητήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να φροντίσουμε αυτές οι μικρομεσαίες να καλυφθούν από το κοινωνικό δίκτυο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Αφενός θα γίνουν ορατές και αφετέρου θα, θα τύχουν μεγαλύτερης αναγνώρισης της σημασία τους για αυτό το δίκτυο, των συνεταιρισμών δηλαδή. Πιστεύω ότι, δηλαδή γενικά ε, συμφωνώ με αυτά τα οποία λες, δεν είμαι σκιώδης εισηγητής, αλλά πιστεύω ότι το θέμα αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, και, και ανοίγει τις πόρτες για μια μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον αντιπρόσωπο της Κομισιόν κύριο Απόστολο Ιακημίδη. Thank you, Chairman. We should like I come from DG Enterprise. Ευχαριστώ. Προέρχομαι από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων που έχει μία διεύθυνση υπεύθυνη για αμοιβέ εταιρείε και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, και για τον συγητή για την έκθεσή του αυτή η οποία ε, περιλαμβάνει πάρα πολλές προκλήσεις ε, επικρίνει στεναρά την Κομισιόν και έτσι μας δίνει την ευκαιρία να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα σχόλια την ε, ε, επόμενη έκθεση την οποία θα υποβάλουμε μέσα στη διαδικασία της συνέχισης. Ε, όσον αφορά τώρα τους συνεταιρισμούς και βάση των στατιστικών στοιχείων, έχουμε στην Ευρώπη 232.000 συνεταιρισμούς αλλά μόνο 17 ευρωπαϊκού μοντέλου. Εάν λάβουμε υπόψη ότι στις κεφαλουχικές εταιρείες. Έχουμε πάνω από 50 εκατομμύρια ιδιωτικέ και δημόσιες εταιρείες και μόνο 600-700 ε, ευρωπαϊκές εταιρείες. Καταλαβαίνετε πόσο επιτυχές, ε, πόσο επιτυχής, ε, επιτυχές είναι το καθεστώς των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών, καθαρά από στατιστικής άποψης και μαθηματικών στοιχείων ο εισηγητής. Κοιτάξτε, εγώ είμαι οικονομολόγος και έχω κάποιο υπόβαθρο στα μαθηματικά. Παρόλο που αυτού του είδους τα υψηλά μαθηματικά είναι λίγο άπιαστα για μένα σα ε, σας ευχαριστώ που ε, υποστηρίζετε, την, που διαβάσατε την έκθεση και που είπατε ότι θα απαντήσετε. Όμως δεν συγκρίνεται τον αριθμό των εργαζομένων και εκεί υπάρχουν οι υπό τις διάφορες νομικές μορφές, ε, νομικό καθεστώς. Για 32 ανθρώπους μιλάμε από αυτές τις 17 ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις. Είπα λοιπόν ότι ο ρυθμός των νομικών συμβούλων που εργάζονται μέσα στο πλαίσιο αυτών των 17 είναι πολύ μεγαλύτερος από τους καθεαυτό εργαζόμενους και από τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν. Γι' αυτό ε, συνάγω από τα από σχόλια που άκουσα ότι συμφωνείτε με αυτή την ε, ε, μη ικανοποιητική κατάσταση. Προφανώς το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού δεν είχε στόχο ότι όλοι οι συνεταιρισμοί που χρησιμοποιούσαν την κοινή αγορά θα πρέπει τώρα να μεταβούν σε μια ευρωπαϊκή νομική μορφή λειτουργίας. Βεβαίω, ένα συνεταιρισμό όπως κάθε άλλη επιχειρήση έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί διακρατικά ή διασυνοριακά χωρί να χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή νομική μορφή. Υπάρχουν συνεταιρισμοί σε πάρα πολλέ ε, χώρες και όταν συνεργάζονται πρέπει να έχουν ένα νομικό καθεστώ λειτουργία, το οποίο προσαρμόζεται στις συγκεκριμένε του ανάγκε. Ε, υπάρχουν ιδιαιτερότητες συνεργασίας. Και αυτές, αυτοί οι συνεταιρισμοί που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας λένε ότι υπάρχουν προβλήματα με το καταστατικό λειτουργίας τα οποία πρέπει να λυθούν. Άρα μας στέλνουν ένα μήνυμα ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και βέβαια συμμερίζουμε την άποψή σας ότι το να απαλλαχθούμε από τη γραφειοκρατία δεν είναι αυτός σκοπός. Βεβαίως υπάρχει ανάγκη κανονισμών ενός κανονιστικού πλαισίου και αυτό το πλαίσιο πρέπει να φροντίσει για την ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, την, απο, την καταπολέμηση των απατών, ε, την αύξηση της αξιοπιστίας μεταξύ οικονομικών εταίρων και λοιπά. Όλα αυτά τα καλά να γίνουν με το ελάχιστο της γραφειοκρατίας χωρίς όμως να ε, διαταράξουμε ε, τους οικονομικά συνεργαζόμενους αν δεν υπάρχει ανάγκη. Οι εταίροι και οι συνεργάτες δεν πρέπει να διαταραχθούν. Δεν θέλω να ερμηνευθεί αυτή η πρόταση ότι είναι ε, μια, μια, μια πρόφαση για, την, για, για προσκόμματα στην εργασία. Και εγώ είμαι μέλος στη συνεταιριστική μου ε, ε, τράπεζα και πολλές φορές με αποκαλούν σύντροφο, πράγμα στο οποίο είναι συνηθισμένο, είμαι συνηθισμένος εγώ από το κόμμα των Πρασίνων, ιδίως η Γερμανία. Πιστεύω ότι εάν είχαμε ενισχύσει των συνεστικών τραπεζών θα είχαμε τώρα πολύ λιγότερα προβλήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε. Πολλές φορές βεβαίως έχει γίνει και καταχρηστική χρήση της έννοιας του συνεταιρισμού. Καμία σωστή ιδέα παγκοσμίω δεν έχει τύχει καταχρηστικής ερμηνείας πολλά πράγματα, καλά πράγματα έχουν, ε, σε αυτά έχουν γίνει καταχρήσεις. Επίσης το παράδειγμα όπου μια ιδέα ενό συνεταιρισμού που υποτίθεται ότι υπηρετεί το κοινό καλό και τις ε, κοινωνικές, το, το κοινωνικό αγαθό έχει, έχει χαθεί. Έχει χαθεί, δηλαδή ορισμένοι συνεταιρισμοί ξέχασαν την, τον ηθικό τους στόχο και λειτουργούν σαν ε, κερδοσκοπικές οργανώσεις με όλα τα δεινά, ας πούμε, άλλων μεγάλων επιχειρήσεων ε, ως αρπακτικά, αρπακτικές εταιρείες. Είπε και η Νάντια Χίρς, η κυρία Χίρς, και αν προφέρεται η κυρία Χίρς πολύ διαφορετικά από ό,τι ε, θα έπρεπε στη γερμανική γλώσσα, ε, Υπάρχει ανάγκη λοιπόν υποστήριξης του τομέα και αναγνώρισης ε, των, ε, των κοινωνικών ωφελών που μπορεί να προσφέρει. Ο, πρέπει όμως να τα κάνουμε όλα αυτά χωρίς να ε, πιστεύουμε, χωρίς να δηλώνουμε ότι όλα είναι πολύ καλά και ωραία μπορούμε να διορθώσουμε τα κακό κείμενα με τον κατάλογο των προτάσεων που έχουμε υποβάλει και που, θα εξετάσει το Κοινοβούλιο. Ε, προσβλέπω λοιπόν ε, σε μια επικοδομητική συνεργασία και θα μελετήσω τις τροπολογίες σας. Ε, έχει ε, αλλάξει η ημερομηνία υποβολή τη έκθεση. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για τι τροπολογίε. Είμαστε πιεσμένοι από χρόνο. Παρακαλώ, υποβάλτε τι τροπολογίε για να οργανώσω εγώ μετά τι σκιώδει διαβουλεύσει και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε απαντώντα τι συστάσει τη Κομισιόν. Και είμαι βέβαιο ότι κάτι καλό θα προκύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, με συγχωρείτε για το όνομα, δεν ξέρω αν είναι κυρία Ιχς ε, κάποιος θα πρέπει να μου εξηγήσει τη ε, διαφορά. Θα ήθελα πολύ να μάθω να αποκτήσω μία μόνιμη εκπαίδευση σε αυτό το θέμα. Έχουμε ολοκληρώσει αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης για το οποίο δίνουμε πολύ μικρή προθεσμία υποβολή ε, τροπολογιών για αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, στι 7 Νοεμβρίου και να συντάξουμε το συμβιβαστικό κείμενο για τις 22 Νοεμβρίου και να το εγκρίνουμε 23 Νοεμβρίου. Περνάμε στο πρώτο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης, το σημείο 15 θα δώσω το λόγο στην κυρία Καρυμαντέλη για την εξέταση των τροπολογιών όσον αφορά την εκθεσή τη για την ενδιάμεση αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2007-2012 σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των τροπολογιών. Έλαβα πάνω από 240 τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις συζητητές και όσους δεν ήταν σκιώδεις συζητητές επίσης και που μας υπέβαλαν τις δικές τους τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κοιτώντας το σύνολο των τροπολογιών προκύπτουν πολλοί συμβιβασμοί για πολύ σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο που αφορά την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων, το είδαμε σήμερα το πρωί με την ακρόαση για το στρες στο χώρο εργασίας και αυτό το κομμάτι θα αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού, τουλάχιστον ελπίζω, ενό συμβιβασμού που θα μας υπενθυμίσει την κοινή υπευθυνότητα και αλληλέγγυη υπευθυνότητα όλων τον κρίκο της αλυσίδας που εργάζονται στην υπεργολαβία. Στοιχείο κλειδί αυτής της έκθεσης. Συμβιβασμός λοιπόν που ε, προσβλέπει προς την προστασία, προστασία και που λαμβάνει υπόψη τις διαφορές, τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και όσα αφορούν τα άτομα με αναπηρίες και κυρίως όσους ε, έχουν αναπηρίες ε, που διαφέρονται εντονότερα στο χώρο εργασίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη μελέτη των τροπολογιών. Θα προτείνω τον πρώτο συμβιβασμό πριν από τις 12 Οκτωβρίου, πριν την επόμενη εβδομάδα και θα αρχίσουμε πραγματικά να έχουμε συνεδριάσεις σκιωδών εισηγητών ώστε πολύ γρήγορα να, ε, συμπερα... να καταλήξουμε σε συμβιβασμού και να είμαστε σίγουροι ότι η έκθεση θα βρίσκεται στο ύψο των προκλήσεων, της πρόκλησης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόκληση. Η υγεία στο χώρο εργασίας, πρέπει να το υπονθυμίσουμε, είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν τη διασφάλιση, τη νομική διασφάλιση συνθήκων εργασίας που σέβονται την υγεία, την ασφάλεια αλλά και κυρίως την αξιοπρέπειά του. Το έχουμε αντιληφθεί σε πολλές ακροάσεις που διεξήγαμε ότι σήμερα διαπιστώνουμε, πιστεύω όλοι μας, ε, είμαι πεπισμένοι. ωστόσο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και πολύ περισσότερο. Σας υπενθυμίζω, η έκθεση μου πρέπει να βγει από την Επιτροπή Απασχόλησης με κυρίως νομοθετικούς περιορισμούς με τρόπο λειτουργίας, με ένα μήνυμα το να σταματήσουμε τα προβλήματα στην εργασία, να υπενθυμίσουμε όλες τις πολιτικές που πρέπει να υλοποιήσουμε και όλες τις επαγγελματικές ασθένειες που διαφαίνονται και που δεν έχουν πραγματικά ληφθεί υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μιλώ κυρίως για τους καρκίνους που προκύπτουν από τους χώρους εργασίας, τις ε, νέες τεχνολογίες, ε, αυτό το άνοιγμα της οδηγίας REACH, με τους χημικούς και βιολογικούς κινδύνους και ο δεσμευτικός, να υπάρχει ο δεσμευτικός στόχος που θα μας την, ότι οι επιθεωρητές εργασίες που σήμερα πρέπει σήμερα οπωσδήποτε να αναγνωριστούν, να αξιοποιούνται και να είναι παρόντες στις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν υπάρχει αυτή η πρόκληση για τις συνθήκες εργασίας. Τώρα απαιτείται πολιτική βούληση και πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά πολύ γρήγορα. Περιμένω λοιπόν ε, τις συνεδριάσεις ε, με ανυπομονησία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχουν εγγραφεί τρεις ομιλητές. Κλείνω τη λίστα των ομιλητών. Η κυρία Ράπτη, ο κύριος Μπακ και ο κύριος Κρίστενσεν. Κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, και μετά από εσά να ευχαριστήσω την Καρίμα η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά, μας προσέφερε ένα εξαιρετικό κείμενο βάσης για να εργαστούμε. Έχουμε κάνει και ως σοσιαλιστές και εγώ προσωπικά ε, κάποιες τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο πνεύμα με την εισήγηση που έκανε η Καρή Ντελή και ε, πραγματικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για την επίτευξη συμβιβασμών. Ε, θέλω να πω μερικά πράγματα ε, που ε, λένε, δείχνουν το πού κινούνται οι τροπολογίες μας και το πνεύμα, και το πνεύμα μας. Ε, θέλουμε σωστές, οι σωστές συνθήκες εργασίας να είναι κριτήριο για την ανάθεση έργων σε επιχειρήσεις, ώστε να ανταμείβονται οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες που λειτουργούν με πολιτικές κοινωνικής ευθύνης. Ε, θέλουμε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η πολιτική πρόληψης μέσω της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εργασίας. Έχουμε στο μυαλό μας περαιτέρω έρευνα να γίνει για να εντοπίζονται οι νέοι κίνδυνοι, οι καινούργιοι κίνδυνοι στην εργασία από τα καινούργια υλικά που χρησιμοποιούνται και βεβαίως να αξιολογούνται επακέλματα τα οποία μέχρι τώρα δεν τα θεωρούσαμε επικίνδυνα αλλά προκύπτει τώρα η επικινδυνότητά τους ε, υπερθεματίζουμε και στηρίζουμε την πρόταση της εισηγήτριας για μια οδηγία που αφορά το στρες στην εργασία και ζητάμε πολύ σοβαρή έρευνα στο φαινόμενο των αυτοκτονιών που παρατηρούνται όλο και συχνότερα και δυστυχώς ε, συνδέονται με το εργασιακό στρες. Και εδώ να τονίσω ότι αυτή η ενημέρωση που είχαμε το πρωί την παρακολουθούσα από το γραφείο μου γιατί έπρεπε να ετοιμαστώ για μια ε, άλλη έκθεση στην ΙΜΚΟ για το στρες ήταν πραγματικά φοβερή και εξαιρετική ταυτοχρόνως. Ε, ειδική μέρημνα για τις ευάλωτες ομάδες εργαζομένων, ε, καλύτερη χρήση των στατιστικών στοιχείων και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών. Αυτό που είπε και η Καρίμα για το θέμα των επιθεωρητών εργασίας, συχνότερη αποτελεσματική έλεγχη ώστε να αξιολογούνται πραγματικά οι κίνδυνοι, να προστατεύουμε όσους καταγγέλουν παράνομες ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και ε, να δώσουμε βάση και ειδική φροντίδα και μέρημνα στους εργαζόμενους οι οποίοι επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από κάποιο ατύχημα ή μετά από κάποια ασθένεια. Τέλος, ε, νομίζω ότι οι τιμές και οι δείκτες που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία έχει σημασία καθώς απλοποιούμε την νομοθεσία μας, να μην πηγαίνουν πιο κάτω. Πρέπει να διατηρούνται στα σωστά επίπεδα. Βάζω μια τελεία. Ευχαριστώ και πάλι την Καρίμα και νομίζω ότι θα έχουμε εξαιρετική συνεργασία όπως και μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καρή Μαντέλη για την εξαιρετική της εργασία. Το πρώτο προσχέδιο ήταν πολύ συγκεκριμένο, είχε απτό περιεχόμενο και νομίζω ότι με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να προσθέσουμε ορισμένες ε, τροπολογίες για συμπλήρωση της έκθεσης. Ως προς το περιεχόμενο θεωρώ ότι ότι δεν υπάρχουν ε, μεγάλες αποκλίσεις απόψεων. Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο στα εξής. Θα θέλαμε να υπάρχει ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των διαφόρων φορέων, δηλαδή να επενδύσουμε σε προληπτικές δράσεις ιδιαίτερα και να είναι, όπου να είναι κοινωνός άμεσα ο εργαζόμενος ως προς την υπεργολαβία Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μείζον πρόβλημα, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν αλυσιδωτές υπεργολαβίες και εδώ υπάρχει μεγάλη επισφάλεια ως προς το μισθό των εργαζαμένων. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους και τις κυρώσεις δηλαδή τα ε, ανθρώπινα μέσα και τις επιθεωρήσεις, να έχουμε, μεγαλύτε, να έχουμε περισσότερους, με συγχωρείτε, επιθεωρητές εργασίες, εργασίας. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους whistleblowers, αυτούς που κοινοποιούν τα κακό κείμενα στην επιχείρηση, για να δούμε ε, πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα υγείας και να δούμε τις πρακτικές στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, ίσως διχογνωμίες που θα φανούν τις επόμενες μέρες ως προς το θέμα της νομοθεσίας, δηλαδή πώς μπορούμε να νομοθετήσουμε καλύτερα και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε καλύτερα την υπάρχουσα νομοθεσία. Το είπε και η εισηγήτρια αυτό, ότι χρειαζόμαστε επιπρόσθετα νομοθετικά μέσα. Ιδιαίτερα για τις αλυσιδωτές υπεργολαβίες και θα πρέπει να, να υπάρχει μια νομοθεσία ως προς το άγχος στην εργασία. Είμαι σίγουρος ότι η συγγήτρια θα βρει πολύ καλούς συμβιβασμούς και χαίρομαι εκ των προτέρων γι' αυτό. Ο κύριος σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ επίσης και την κυρία Ντέλη για όλη αυτή την πολλή δουλειά που έκανε για αυτή την έκθεση μέχρι τώρα. Δύο σημεία θα ήθελα να αναφέρω που είναι πολύ συγκεκριμένα και εξειδικευμένα. Έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες με την Σιλβάνα Ράπτη από κοινού. Η Σιλβάνα είναι η δική μας ε, σκιώδηση συγγήτρια για αυτό το θέμα. Είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα αυτό το οποίο ε, έχει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ο αμύαντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα στην υγεία και ασφάλεια που θέτει ο αμύαντος. Ο αμύαντος στα κτίρια, στα πλοία, στα τρένα, σε, στον μηχανολογικό εξοπλισμό είναι μεγάλος κίνδυνος. Άνθρωποι πεθαίνουν λόγω του ότι εκτίθενται και έρχονται σε επαφή με τον αμίαντο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξει πρόγραμμα ώστε τα κράτη-μέλη να πάψουν να χρησιμοποιούν, όχι μόνο να πάψουν να χρησιμοποιούν, αλλά η απαγόρευση της χρήσης του αμίαντου να δώσει λύσεις. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι θα δοθούν λύσεις και θα υπάρχουν κανόνες ασφάλειας για την αφαίρεση και από ε, ξύλωση ε, ε, αμοιάντου υπάρχει ένα ευρύτατο, ένα, ε, ένα, ένα ευρύ φάσμα που δεν έχει ληφθεί υπόψη και συμπεριλαμβάνει τομείς και παιδεία όπου θα ε, μου γνωστοποιήθηκαν και συνειδητοποιήσαμε υπάρχει έλλειψη κανόνων και κανονισμών. Χρειάζεται άμεση δυνατότητα δραστηριοποίησης. Όσον αφορά για παράδειγμα τις κομμότριες, ε, οι κομμότριες ε, και οι κομμωτές εργάζονται με χημικά προϊόντα τα οποία είναι και επικίνδυνα. Και αν δει κανείς για παράδειγμα τη χρονική στιγμή συγκυρία και την απασχόληση αυτών των, το χρόνο απασχόλησης ε, των κομμωτών ε, και κομμωτριών είναι μικρός ε, διότι ασθενούν συχνά τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, σε σχέση και με τους ε, πιλότους ε, δεν θα πρέπει να εκτίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν και κίνδυνοι από ατυχήματα. Υπάρχουν σωματίδια, πολύ μικρά ε, σωματίδια τα οποία είναι, προξενούν καρκίνο, είναι καρκινογόνα. Είναι ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό για όσους εργάζονται σε τέτοιους χώρους και προσβάλλονται με αυτό, εκτίθενται και προσβάλλονται έτσι. Επίσης υπάρχει και το θέμα των ε, όσων ε, χειρίζονται αποσκευές ε, και ξεφορτώνουν, φορτώνουν και ρυθμίζουν τα θέματα αποσκευών ε, εκτίθενται και αυτοί όσον αφορά. Και όσον αφορά επίσης άλλο θέμα, ε, η χρόνια οδήγηση ε, δεν εφαρμόζονται σε σχέση με οδηγούς λεωφορείων που καλύπτουν αποστάσεις μικρότερες από 50 χιλιόμετρα διαμιάς σε μια περίοδο δραστηριοποίησης. Είναι λοιπόν σημαντικά μηνύματα να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Κυρία Ντέλη, παρακαλώ, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους σκιώδεις και τους ε, βουλευτές ε, για αυτά τα στοιχεία ως προς τις τροπολογίες. Τι? Βεβαίως θα πρέπει να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πολιτικές υγείας. Θα πρέπει να τις συσχετίσουμε με όλες τις άλλες δημόσιες πολιτικές, δηλαδή απασχόληση, μεταφορές, ενέργεια, κατάρτιση, περιβάλλον, κλιματικές αλλαγές και ούτω το καθεξής. Είπατε πολύ σωστά κύριε Κρίστεσεν ότι θα πρέπει να, να αντισταθούμε στην τοξικότητα και στους νέους χημικούς και βιολογικούς κινδύνους. Μιλήσατε για το REACH και για τον αμίαντο. Θα πρέπει να ξανανοίξει αυτή η οδηγία REACH. κάτι το οποίο διαφαίνεται και από την έκθεση. Συμφωνώ και με το θέμα της υπεργολαβίας για μένα θα πρέπει να αποτελέσει επίκεντρο το, της γνωμοδότησής μας, γιατί μπορούμε να φτάσουμε σε υπεργολοβία σε επίπεδο μείον 8. Δηλαδή μιλάμε για αλυσιδωτές υπεργολαβίες. Και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, επανοργανώσουμε τον εργασιακό χώρο. Χαίρομαι διότι φύγεται το, το θέμα των κοινοποιητών ε, δυσλειτουργιών, των whistleblowers, γιατί πολλές φορές μιλάνε για θέματα διαχείρισης κινδύνων και πολλές φορές δεν προστατεύονται, ίσα ίσα απομακρύνονται. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη, το είπατε, και σε σχέση με το επίπεδο κυρώσεων θα πρέπει να το δούμε στο σύνολο της έκθεσης. Θα πρέπει να φτάσουμε σε συμβιβασμούς, ορόσημα, έτσι ώστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αποφανθεί το Κοινοβούλιο επί του θέματος ολοκληρωτικά. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Μου ανέφεραν ότι ο Επίτροπος θα μιλήσει στον τύπο πριν ε, προσέλθει. Άρα θα περιμένουμε μερικά λεπτά, μη φύγετε όλοι και όλες, ας κάνουμε μία μικρή διακοπή για να τον περιμένουμε. Πριν όμως, πριν όμως, λέει η Πρόεδρος, ξέχασα ως προς σημείο 15 να σας αναφέρω τα εξής. Ε, αν λάβουμε υπόψη και αυτό το βήμα που διανύσαμε, θα ξανασυναντηθούμε στις 7 Νοεμβρίου για να συζητήσουμε τις τροπολογίες συμβιβασμού πριν ψηφιστούν στις 23 Νοεμβρίου. Τελειώσαμε και με το 15 και διακόπτουμε για λίγα λεπτά, ε, κάνοντας με την παράκληση να μην απομακρυνθείτε. Chers Σας προτείνω να... συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Έχουμε ακριβώς μισή ώρα. Ο Επίτροπος θα μας παρουσιάσει τις προτάσεις που υιοθετήθηκαν και αφορούν τη συνολική δομή για τα διαφορετικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Του δίνω το λόγο χωρίς καθυστέρηση. Μας ήρθε από μια press conference. Ε, έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Uh, uh, Καλή σας μέρα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά για τα τρία έγγραφα για τα οποία θα σας κάνω λόγο σε 9.30 τα υπέγραψα σήμερα και είχαμε μια πρώτη συνέντευξη με τον Επίτροπο Χάν και πολλά θέματα, ιδιαίτερα γύρω από μια πτυχή του πακέτου που εγκρίθηκε σήμερα και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα οποία θα συζητήσουμε είτε σήμερα είτε και με άλλη ευκαιρία θα θίξουν, θα καλύψουν αυτές τις πτυχές. Ας ξεκινήσω καλύτερα λέγοντας ότι Αυτά τα οποία συζητήθηκαν σήμερα συνδέονται και με τον λόγο του Προέδρου για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγο που εξεφώνησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι όπως είπε η Ευρώπη βρίσκεται σε μια καμπή, σε ένα σταυροδρόμι και είναι σαφές ότι η μελλοντική ανάπτυξη διακυβεύεται Πραγματικά οι προβλέψεις, ε, οι προγνώσεις δείχνουν ότι σε πάρα πολλές χώρες παγκόσμια, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες, πρέπει να δούμε αυτή την προοπτική και δεν αποτελεί εξαίρεση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη είχαμε σε σχέση με τη μείωση του, ε, ε, της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν αυτό το φαινόμενο. Δεύτερο μέλημα είναι η απασχόληση. Σε σχέση με την άνοιξη όπου είχαμε την προοπτική ανάκαμψη, τώρα πρέπει να φοβούμεθα για μια κάμψη με αρνητική φθήνουσα πορεία για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, υψηλότατη διαθροτική ανεργία με πάρα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Υψηλότατη ανεργία σε σχέση με μείωση ανάπτυξης που αποκλείει εργαζόμενους και από την αγορά εργασίας και τους αποκλείει κοινωνικά και τους θέτει στο περιθώριο. Καθώς επίσης και αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης και επισφαλούς διαβίωσης. Αυτή η ε, εξέλιξη σε σχέση με την αύξηση των περιορισμένου χρόνου ε, δυνατοτήτων απασχόλησης, περιορισμένης δηλαδή εργασίας, τρίτον η υψηλότατη ανεργία των νέων, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Η ανεργία των νέων παραμένει υψηλότατη σε διπλάσιο επίπεδο από το επίπεδο ανεργίας των ενηλίκων και αυξανόμενη κοινωνική αναταραχή όσον αφορά την υιοθέτηση αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων περικοπών και λιτότητα στα κράτη-μέλη και όσον αφορά την ε, ανισότητα και τις ε, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις που προκαλούν όλα αυτά. Υπάρχει όλο και αυξημένη αίσθηση στους Ευρωπαίους ότι το κόστος ε, της κρίσης δεν το συμμερίζονται όλοι με τον πιο σωστό δίκαιο τρόπο και το είδαμε αυτό ότι δημιουργεί μια ιδιαίτερα εκρηκτική κατάσταση. Αναθεώρη, ε, μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας καθώς επίσης και άλλες ε, μεταρρυθμίσεις σε σχέση με την ε, λιγότερο αυξημένη ανάπτυξη. Όμως ε, επιτυχία θα επιτευχθεί μόνο αν δημιουργούν, δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Είναι ζωτική σημασία να δοθεί συνέχεια στην παρακολούθηση αυτών των στόχων διαθετικά δίνοντας την ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και δημιουργία διαθέσεων απασχόλησης. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, παρότι οι κύριες ευθύνε για την πολιτική ε, της ε, αγοράς εργασίας είναι των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα από πλευράς δημοσιονομικής από πλευράς προπολογισμού μπορούμε να συνεισφέρουμε. Αυτά τα οποία υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο <clears throat> καθορίζουν το πώς θα μπορέσει ο προπολογισμό να συνεισφέρει να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο στοιχεία εδώ πρέπει να τονιστούν. Η αλληλεγγύη που πρέπει να δημιουργηθεί και ως πλαίσιο να ισχύει για τα φτωχότερα κράτη-μέλη και τις ε, ομάδες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Ε, δεύτερον, ένα μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού θα στοχεύει στο να ξαναενεργοποιηθούν θέσεις απασχόλησης και να συνεισφέρουμε έτσι στην οικονομική αναπτύξη. Και έτσι αυτό αφορά την στρατηγική για μια ε, αποτελεσματικότερη δράση. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να σας πω ότι υιοθέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πολιτική για τη συνοχή και την ανάπτυξη και τις πρώτες προτάσεις ε, όσον αφορά τα πολιτή ε, δημοσιονομικά πλαίσια. Είναι σημαντικό αυτά τα μέσα για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, το ESF, το DGF και το νέο πρόγραμμα για την καινοτομία και την ε, ε, ανάκαμψη αλληλοσυνδέονται στενά και είναι ζωτική σημασία να διασφαλίσουμε την παραπληρωματικότητά τους. Θα ήθελα να δραχθώ τη ευκαιρία σύντομα να αναφερθώ σε αυτά και να τονίσω κάποιες από τις αλλαγές που προτείναμε ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε και να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Να ξεκινήσω με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όπως είχε προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση για τα πολιετή πλαίσια, οι κυριότερε προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα ανταποκρίνονται απόλυτα στην στρατηγική για το 2020. Θα επικεντρώνεται σε τέσσερι τομεί. Απασχόληση και κινητικότητα, κατάρτιση και διαβίου εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση τη φτώχεια και θεσμική δημιουργικότητα και ικανότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω αυτών των προτεραιοτήτων θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, ιδιαίτερα από το 7 έως το 10 και των κυριότερων πρωτοβουλειών, ιδιαίτερα της πλατφόρμας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να ε, τονωθεί αυτή η πτυχή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω τους στόχους που πρέπει ως προτεραιότητα να αντιμετωπιστούν, καταπολέμησης ανεργίας των νέων και ε, βοήθεια στις ε, περιθωριοποιημένες ομάδες, ε, ευάλωτες ομάδες όπως τους Τσιγκάνους, του Ρώμα. Πολλά περισσότερα πρέπει και μπορούν να γίνουν για να προλάβουμε και να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό η πρότασή μου, τουλάχιστον η πρότασή μας, 20% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να προκαθοριστούν για δράση σε αυτή την κατεύθυνση. Πράγματι πρέπει να προαχθεί επίσης και η ισότητα των φύλων και η ισότητα ευκαιριών που πρέπει να είναι κύριοι στόχοι για την δραστηριοποίηση των κονδυλίων του κοινωνικού Κοινωνικού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από τα κράτη-μέλη να επικεντρώσουν τις ε, χρηματοδοτήσεις από τα ταμεία στα θέματα που έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί στα εθνικά προγράμματα και στις συστάσεις ανάλογα με τις χώρες. Αυτό θα ζητεί περαιτέρω προτεραιότητες να λαμβάνονται υπόψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πιο ανεπτυγμένες ε, χώρες τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα είναι ισχνά, θα είναι λιγότερα και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους στόχους. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις και δείκτες επιδόσεων για να κατανέμονται. Αξιότιμα μέλη, μέχρι σήμερα η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον προπολογισμό ήταν αποτέλεσμα διμερών διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη. Κατά τα τελευταία 20 χρόνια το μέρος αυτό από 40% το μερίδιο αυτό κατέληξε περίπου στο 22 20 με 22% όλο και περισσότερο ζητούσαμε να υπάρξουν επενδύσεις ε, για τους ε, ανθρώπους, το ανθρώπινο δυναμικό, την καταπολέμηση της φτώχειας. Είναι μια άποψη που συμμεριζόμαστε όλοι, ότι πρέπει να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ των στόχων, των κοινών συμφερόντων και των πραγματικών δυνατοτήτων κατανομής επιμερισμού κονδυλίων δημοσιονομικά. Στις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν με ιδιαίτερη φροντίδα θα μεριμνήσει η Επιτροπή ώστε επαρκές τμήμα της χρηματοδότησης να προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουμε προτείνει ελάχιστα επίπεδα για κάθε περιοχή και για κάθε κατηγορία. 25% για τις ε, περιοχές σύγκλησης, 40% για τις μεταβατικές περιοχές και 52% για τις περιοχές ανταγωνιστικότητας ανταγωνιστικές περιοχές. Να είναι σαφές αυτό. Δεν είναι μια ισοπεδωτική προσέγγιση με μια πρόταση που θα ισχύει για όλους. Θα διασφαλίζει τα ελάχιστα επίπεδα ώστε να ανταποκρίνονται οι επενδύσεις, η χρηματοδότηση να ανταποκρίνεται με τις ανάγκες. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά επιτόπου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να λειτουργούν καλύτερα και να είναι πιο αποτελεσματικά. Πρέπει να υπάρξουν οι μηχανισμοί στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών και περιφερειών, ώστε να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση στην πολιτική συνοχή. Και θέλουμε εν τέλει ως Επιτροπή να προαγάγουμε την εξαπλούστευση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ιδιαίτερα για τους τελικούς αποδέκτες. Οι προτάσεις θα λαμβάνουν υπόψη αυτές τις προτάσεις και θα τις προαγάγουν. Επιπλέον θα προαγάγουν μεγαλύτερη τυποποίηση και θα βοηθούν ώστε να αρθεί η νομική αβεβαιότητα, η, η ανασφάλεια όσον αφορά τα κρατημέλη. Επίσης ένα κοινό πρόγραμμα δράσης θα συμπεριλαμβάνει ένα μέτρο δράσεων που θα συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληρωμές και οι έλεγχοι θα εξαρτώνται απόλυτα από την ανταπόκριση σε όρους και προϋποθέσεις και συγκεκριμένες ε, διατάξεις και κανονισμούς. Όπως βλέπετε, στοχεύουμε να υλοποιήσουμε μια πρόταση που θα ε, ενδυναμώσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είμαστε πεισμένοι ως Επιτροπή ότι είναι η μόνη πορεία που μπορεί να ακολουθηθεί αν θέλουμε αξιόπιστα να συνεισφέρουμε στην ανταγωνιστικότητα και ανάκαμψη με δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η επιτυχία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την χρήση και τις ευκαιρίες που θα δοθούν μέσω αυτών. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, το δεύτερο μέσο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω σε εσά είναι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Στοιχείο που έχει σημασία κλειδιού και θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργήσει και στο μέλλον καταδεικνύει το Ταμείο αυτό την αλληλεγγύη με εργαζόμενους που επειδή κατέστησαν περιττή και δεν μπορούσαν να απασχοληθούν, απελήθησαν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους. Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 78 αιτήματα υποστήριξης από το Ταμείο Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση από 9 κράτη-μέλη και για 358 εκατομμύρια ευρώ συνολικά που 76.000 εργαζόμενους ε, θα ε, βοηθούσαν. Επίσης όμως παρόλα αυτά πρέπει να διασφαλίσουμε ώστε να μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση και στο μέλλον. Ο μηχανισμός πυρήνας ε, του, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα διατηρηθεί και θα συνεχίσει έτσι να λειτουργεί όσον αφορά τους εργαζόμενους που κατέστησαν άνεργοι θα έχουμε και την συγκεκριμένη προθεσμία για την υλοποίηση αυτών των μέτρων. Επιπλέον όμως θα παραμείνει εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μέγιστο ποσό κατά τη θα μειωθεί σε 430 εκατομμύρια. Και γι' αυτό υπάρχουν και τέσσερα νέα στοιχεία όσον αφορά τον κανονισμό του Ταμείου αυτού. Θα προτείνουμε την διεύνηση σε νέες κατηγορίες εργαζομένων που αυτή τη στιγμή ε, εξαιρούνται δυστυχώς ε, στην πρακτική εφαρμογή. Για παράδειγμα, προσωρινά εργαζόμενους ή εργαζόμενους με συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας, αυτοαπασχολούμενους, ε, καθώς επίσης και όσον αφορά και τα ταμεία για τις δράσεις για τους μικρομεσαίους. Επίσης, οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες που θα συναυθούν από την Ένωση ε, θα λάβουν υπόψη το στόχο και το πεδίο ενισχύ ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην ε, παγκοσμιοποίηση. Το ταμείο αυτό ταυτόχρονα θα υποστηρίξει οι εργαζόμενους που έχουν χάσει την εργασία του λόγω μιας αναπάντεχης οικονομικής κρίσης η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο και στοπικά τοπικά εργαζόμενους η συγχρηματοδότηση του Ταμείου Προσαρμογής θα συμπεριλάβει 50% χρηματοδότηση του κόστους του πακέτου και των εφαρμοστικών μέτρων, όμως αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί σε 65% σε κράτη-μέλη τα οποία εμπίπτουν στα πεδία σύγκλησης υπό το κοινωνικό ταμείο. Έτσι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε περισσότερους εργαζόμενους με την ίδια ε, με το ίδιο κομμάτι της πίτας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ε, βασιζόμενη στην αλληλεγγύη, στο, στοιχείο της αλληλεγγύης. Και τέλος, θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, θα ζητούμε περισσότερες πληροφορίες στην υποβελή αιτήσεων από τα κράτη-μέλη και θα εφαρμόσουμε κάθε δυνατό μέτρο για να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Επίσης, τρεις μήνες θα είναι το όριο ε, διαχείρισης των ε, εξέτασης των ετοιμάτων ε, και αυτοί οι τρεις μήνες ε, θα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής ε, της αίτησης μέχρι την υποβολή καταβολή των πιστώσεων. Επίσης η Κομισιόν θα υποβάλει ένα καινούριο πρόγραμμα για κοινωνικές αλλαγές και καινοτομίες, το οποίο θα συμπληρώνει άλλα μέσα όπου όπως το ESF και το EGF, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ο προϋπολογισμός ε, θα καλύπτει το μέσον αυτό με 500 εκατομμύρια. ευρώ και θα δώσει επίσης τη δυνατότητα εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας το, η χρηματοδότηση αυτή θα διευκολύνει την πρόθεση της ευρωπαϊκής καινοτομίας και, και ιδίως στο κοινωνικό πεδίο. Όταν χρειάζεται κοινωνική παρέμβαση είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό καινοτομικές λύσεις. Μια κοινωνική παρέμβαση απαιτεί καινοτομικέ λύσεις. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να βρουν εργασία στο εξωτερικό σε, σε άλλες χώρες με την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Ήδη το Κοινωνικό Ταμείο ε, παρέχει πληροφορίες ε, για τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας πάνω από 1,2 χαμένες ε, θέσεις εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις τους, υπήρχαν και νέες θέσεις και πάνω από 700.000 βιογραφικά υποβλήθηκαν προς εξέταση. Ε, μέσω του προγράμματος Euros ε, χιλιάδες εργαζόμενοι λαμβάνουν προσφορές εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν το, τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν ε, έναν καλύτερο συγκερασμό μεταξύ υποβολής αιτήσεων και εξέβρισης θέσεων εργασίας. Θα ενισχυθούν επίσης οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει ή δεν μπορούν να βρουν δουλειά με 5.000 ε, ε, επιδοτούμενες σχέσεις εργασίας και θα ε, παρέχει βοήθεια σε μικροχρηματοδοτική κλίμακα για νέες πρωτοβουλίες ή νέες επιχειρήσεις ε, ε, που προσλαμβάνουν άνεργους νέους ή για νέους που, που, θέλουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Έχουμε υπογράψει με 7 κράτη-μέλη ε, συμφωνίες για τη μικροχρηματοδότηση αυτή και άλλες πέντε προβλέπονται μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου. Ως αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών εκατοντάδες επιχειρηματίες έχουν ήδη ενισχυθεί. 420 με 450 εκατομμύρια θα διατηθούν για αυτό το σκαπό. Ε, επίσης ε, θα υποστηρίξουμε ε, το δυναμικό αυτών των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από την μικροχρηματοδότηση. Τα οι προτάσεις αυτές ε, προέκυψαν μετά από καρποφόρες συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβάνουν και το Κοινοβουλίου. Ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, ε, τα παθήματα έγιναν μαθήματα και γι' αυτό πιστεύουμε ότι υποβάλλουμε τις καλύτερες δυνατόν προτάσεις με τις παρούσες συνθήκες Προσβλέπω στις δικές σας, ε, στο να μελετήσω τις δικές σας απόψεις και ιδέες και πιστεύω ότι μπορώ να υπολογίσω στην στήριξη των προσπαθειών μας από αυτή την Επιτροπή έτσι ώστε όλα τα καλά στοιχεία αυτής της πρότασης να περάσουν. Ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε. Ο Επίτροπος ε, δυστυχώς ε, ήρθε με μισή ώρα καθυστέρηση και μας μένουν μόνο δέκα λεπτά. Θα, ίσως θα μπορούσαμε να μείνουμε μέχρι τις μία και τέταρτο, αλλά θα περιορίσω τις ομιλίες σε δύο λεπτά. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρή και μετά στον κύριο Σαρκάς. Σαρκάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα μόνο, γιατί πρόκειται για ένα πρώτο γύρο σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και πρέπει φυσικά να δούμε εξειδικευμένα τι θα εμπεριέχει αυτή η πρόταση. Είδα κάποιες συγκεκριμένες αντιφάσεις ε, από τα όσα ακούσαμε και θα ήθελα να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με αυτά τα θέματα. Στο, στην πολιτική συνοχή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα έπρεπε να διαδραματίζει ένα ευρύτερο, πιο σημαντικό ρόλο. Πολύ καλά. Αλλά από πλευρά Επίτροπή ε, βλέπετε και την άλλη πλευρά. Σκέφτεστε για παράδειγμα και την Ουγγαρία. Καλή ιδέα θα ήταν να δαπανώνται λιγότερα κονδύλια στην δημιουργία νέων πλατιών και να δίνεται μεγαλύτερη που τα μεγαλύτερη προσοχή και σημασία στην δημιουργία θέσεων απασχόληση. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω είναι ένα κανόνα για να υπάρξουν βελτιώσει όσον αφορά το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Το να διευρυνθεί το εύρο, το φάσμα δράσεών του, θα μπορούσε να είναι αρκετά επικίνδυνο να εγκυμονούν κάποιοι κίνδυνοι, ακόμα και αν δεν έχουν ε, όλα τα κονδύλια δαπανηθεί, πολύ σύντομα μπορούν να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού, οι όροι του παιχνιδιού και πολλά θα μπορούσαν να χρειαστούν και να δαπανηθούν πολύ σήμες, άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τι θα κάναμε λοιπόν όταν θα εξαντλούν αυτά τα κονδύλια. Αφορούν τώρα κάτι που αφορά την πρόοδο. Ίσως δεν θα ήταν κακή ιδέα να είχαμε μια πιο θεματολογική, πιο εξειδικευμένη θεματολογικά προσέγγιση εξετάζοντας για παράδειγμα τη νέα προτεραιότητα για την απασχόληση. Πολύ καλή ιδέα αυτή, αλλά με μεγαλύτερη σαφήνεια θα έπρεπε να επικεντρωθούμε σε κάποιους τομείς όπου θα έπρεπε να έχουμε κάποια κατεκτήμηση στοιχεία όσον αφορά την έλλειψη εργατικού δυναμικού ανάλογα με ηλικία ειδικότητα και να μετά να προετοιμαστούν για τέτοιου είδους ε, για, για δράσεις ε, που, για εργασίες όπου απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις και προσόντα οι δεξιότητες τους νέους ώστε να καλυφθούν ε, αυτές οι ανάγκες αυτή στενοπώς να αντιμετωπιστεί όσον αφορά την μικροχρηματική χρηματοδότηση, είναι προς το κοινό συμφέρον φυσικά να στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Και καθώς ελπίζουμε, ελπίζουμε θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες και όταν θα έχουμε διαβάσει όλα αυτά τα στοιχεία και θα έχουμε εξοικειωθεί θα μπορούμε να επανέλθουμε. Αυτά είναι συντομία ευχαριστώ. Ο κύριος Θέρκας, δύο λεπτά, μετά η κυρία Χάρκιν. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Ελπίζω επειδή αξίζει κάτι παραπάνω από δύο λεπτά, να έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε για κάθε μια και για όλα τα ε, κάθε μια από τις πτυχές και όλα τα θέματα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο ανησυχητικό. Πολύ ανησυχητικό γιατί δεν βρισκόταν ούτε στη δική σας παρέμβαση, ούτε στις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που προαναγγέλλονται σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και όμως είναι μια σημαντική τεχνική αλλαγή. Είναι οι όροι και προϋποθέσεις των κονδυλίων αυτού του Ταμείου για την οικονομική κατάσταση των ε, χωρών μας. Η επαναστατική αλλαγή είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο μέλλον Παρόμοια όπως συνέβαινε προηγούμενα με το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορεί να παγώσει και να μην δίνει κονδύλια σε εκείνες τις χώρες που δεν θα υλοποιούν τους οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις ε, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για τους αποδέκτες ε, των κονδυλίων, για εκείνους που θα αποκλείονται από την κοινωνία. Ε, ε, εδώ υπάρχει μια αντίφαση και μια τεράστια στρέβλωση, κύριε Επίτροπε όχι μόνο η κοινωνική ε, ρήτρα δεν εισάγεται, αλλά υπάρχει η μακροοικονομική οριζόντια ε, ρήτρα και η πολιτική εξυπηρετεί την μακροοικονομία και όχι η μακροοικονομία ε, να υπηρετεί την κοινωνία και την κοινωνική συνοχή. Αυτό θα δημιουργήσει και είναι βέβαιο, θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Και λυπούμε πολύ κύριε Επίτροπε να σας πω ότι δημιουργεί και τεράστια προβλήματα για την δική μου πολιτική ομάδα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο σχόλια. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Φέρκα σε σχέση με την αιρεσιμότητα, σε σχέση με το μάκρο και μικροοικονομικό πλαίσιο. Επίσης, βλέπω ότι το Ταμείο Αντιμετώπισης της παγκομιοποίησης θα ασχοληθεί και με θέματα ε, συνοχής. Θα ήθελα να αναφερθώ στα σχόλιά σας ως προς το Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, το EGF. Ποιοι μπορούν να ευεργετηθούν από αυτό. Μιλήσατε και για τους αγρότες που θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση στο Ταμείο αυτό αλλά μιλήσατε και για εμπορικές συμφωνίες ε, στην ίδια σας πρόταση. Υπάρχει συνοχή, δηλαδή εξαιτία εμπορικών συμφωνιών, αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο EGF, στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και θεωρείται ότι οι όροι πρόσβασης θα ήταν οι ίδιοι όπως ισχύει για άλλους εργαζόμενους. Ως προς την μείζωνα κρίση, ξέρω τι έχετε κατά νου, αλλά δεν θα, έπρεπε, δεν θα έπρεπε να υπάρξει αμφισημία, διότι η συγχρηματοδότηση πάντα θα αποτελεί πρόβλημα. Χτες είδαμε την πρώτη αίτηση της Ελλάδας, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η συγχρηματοδότηση μπλοκάρει άλλες χώρες για το EGF. Μιλήσατε για ένα 65% μέχρι το 65%. Μερικοί όμως θα το υπερβούν. Είσαστε ικανοποιημένος με την ε, τρίμηνη προθεσμία και θεωρείτε ότι υπάρχουν ε, στοιχεία του EGF που θα ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να ζητήσουν συγχρηματοδότηση. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να το συζητήσουμε. Η κυρία Σρότερ. Η κυρία Σόρτερ παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ίδια θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι βλέπω ότι υπάρχει λόγος για αυτή την ε, νέα τοποθέτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα θαραλέα αυτά μέτρα και προτάσεις που έχετε παρουσιαστεί θα είναι δύσκολο να τα, να, να τα προασπίσετε. Μπορώ να πω και για την ε, δική μας ομάδα το ίδιο, ότι επειδή θεωρούμε ότι είναι σωστή η κατεύθυνση αυτή. Αυτά τα οποία εμπεριέχονται στη στρατηγική 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορέσουν να επιτευχθούν. Έχουμε και την ουσία και το περιεχόμενο των στόχων αυτών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Είναι τεράστια διεύρυνση του φάσματος δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε σχέση με το παρελθόν. Θα πρέπει να δούμε ότι θα είναι αυτό προ όφελο και κέρδο για τι περιφέρειες και ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο ερωτήσει θα είχα όσον αφορά αυτά. Επειδή δεν είναι απόλυτα σαφέ για τι εννοείται ότι θα γίνει με τη συγχρηματοδότηση. Συγχρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής, με τι χώρε συνοχή με συγχωρείτε. Αυτό τι σημαίνει, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συν το Ταμείο ε, προσαρμογής παγκοσμιοποίησης με αυτόν τον τρόπο θα προαχθούν και θα συγχρηματοδοτούν ή δεν το κατάλαβα καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μωρή Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε μετά από την ε, press conference όπου σας άκουσα με πολύ προσοχή. Θα ήθελα να σας κάνω πέντε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ε, πρώτον, όσον αφορά τις προϋποθέσεις. Θέλουμε να δεσμευτούμε σε μία αρχή διπλής ποινής ε, για τις χώρες που ήδη βρίσκονται, αντιμετωπίζουν οικονομικές και νομισματικές δυσκολίες, ζητώντας τους επιπλέον υπερβολικά ε, μεγάλες συγχρηματοδοτήσεις. Ε, αυτό μας φέρνει και στην παρατηρήση του κ. Σέρκας υπερβολικά βαρύς ε, και δύσκολες για την πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Δεύτερο σημείο, μιλήσατε για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Ο πρώτος μοχλός τον οποίο πρέπει να δράσουμε είναι η καταπολέμηση των πτυχιούχων χωρίς εξειδίκευση. Όσο περισσότερο κάνουμε κάτι τέτοιο πρέπει να περισσότερο θα έχουμε κοινωνικό αποκλεισμό και περισσότερα προγράμματα για την απασχόληση θα πρέπει να δημιουργήσουμε. Στη στρατηγική 2020 πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του και θα πρέπει να κινητοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τους ανειδίκευτους. Το τρίτο σημείο δεν είπατε τίποτα για την ανανέωση των θέσεων εργασίας δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο εξειδίκευσης, το ίδιο επίπεδο απασχόλησης, η φυσιογνωμία, το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας θα αλλάξει από τώρα μέχρι το 2020, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το κοινωνικό ταμείο και για αυτό το στόχο. Δεν μιλήσατε γι' αυτό. Θα παρακολουθούμε στενά την κινητοποίηση του κοινωνικού ταμείου. Το τέταρτο σημείο είναι η κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους γεωργούς. 4.000 ε, που θα έχουν πρόσβαση. Ε, πώς θα γίνει αυτό και το τελευταίο σημείο, κυρία Πρόεδρε, κινητοποίηση του σχεδίου διατροφικής επισητιστικής βοήθειας για τους φτωχότερους, διότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό σε μία ε, ε, ζώνη απολυσίας δικαιωμάτων. Ευχαριστώ για την εισήγηση που κάνατε. Μου δημιουργεί κάποιες ελπίδες, αλλά από την άλλη πλευρά ε, θέλω να ρωτήσω πόσο αισιόδοξο είστε για το κατά πόσον μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά. Και κυρίως, για παράδειγμα, το θέμα των τριών μηνών που θα μεσολαβούν από την αίτηση μέχρι την καταβολή των χρημάτων. Ήταν κάτι που το συζητήσαμε και στην προφορική ερώτηση που είχαν α, καταθέσει η κυρία Μπερές με την κυρία Χάρκιν και συζητήθηκε στο, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ε, ένα ερώτημα που θέλω να κάνω, γιατί από τα, με τα υπόλοιπα καλύφθηκα, είναι το εξής ε, μιλάτε για δημιουργία θέσεων εργασίας. Όταν μιλάμε για δημιουργία θέσεων εργασίας, έχουμε στο μυαλό μας αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας ε, σχετίζονται με τις συνθήκες αλλά και με την αμοιβή. Στην Ελλάδα αυτή την περίοδο και πριν από δύο μέρες αντιμετωπίζουμε αίτημα της Τρόικας και όπως ξέρετε ένα μέρος στην Τρόικα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μειωθεί το ύψος των μισθών στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ε, θα ήθελα ένα σχόλιο, διότι από τη μια μεριά με το ένα χέρι μας δίνεται κάτι και με το άλλο χέρι μας το παίρνετε. Ε, επειδή δε οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι ε, ε ευαγγέλιο για το εργατικό κίνημα, ε, και για μας ποια είναι κόκκινη γραμμή. Θα ήθελα ε, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Α, και κάτι ακόμη. Αντιμετωπίζουμε και το θέμα απολύσεων λόγω της οικονομικής κρίσης στον δημόσιο τομέα. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία και με τον κύριο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Η πρώτη ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης τέθηκε ήδη από την κυρία Χάρκιν η ερώτησή μου και έτσι υποστηρίζω 100% τις δικές της παρατηρήσεις ως προς αυτό. Η δεύτερη μου ερώτηση και αυτή εξίσου καλύφθηκε. Και γι' αυτό η συγκεκριμένη ερώτησή μου προς εμάς κύριε Επίτροπε. Τι έχετε υπόψη να κάνετε με το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για αξιόλογα ποσά και πρέπει να δούμε από πού ε, θα λείπουν αυτά τα κονδύλια, από πού θα αντληθούν και με τη χρήση αυτή ε, από πού θα λείψουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Μάντορα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το βρίσκω ενθαρρυντικό το ότι επισημάνατε πιο πριν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να καταλήξει σε μια απλούστευση. Ένα παράδειγμα, νέες προδιαγραφές και κανονισμοί θα υπάρξουν. Προσδοκώ και αδειμονώ να δω πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, διότι έχουμε σημαντική στοχοθέτηση και ήταν ένα από τα καλύτερα μέσα για να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία η χρήση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και πρέπει να διασφαλιστεί και η διατήρηση αυτής τη αποτελεσματικότητα στο μέλλον. Θέλουμε να, μια και θα είναι μέρος ε, της σύμπραξης για την επίτευξη των στόχων του 2020 να δράσουμε προληπτικά με την αρχή της πρόνοιας και της πρόληψης και όχι μετά να θεραπεύουμε τα κακοσκήμενα. Θα ε, με ικανοποιούσε η καταπολέμηση της ανεργίας ε, των νέων να είναι κύριος στόχος. Πάντα βλέπω να απουσιάζουν σημαντικοί στόχοι από κάποιες χώρες παρότι λέμε ότι θέλουμε να έχουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με αυτό θα πρέπει να βοηθήσει να προχωρήσουμε παραπέρα και να υπάρχουν κίνητρα. Επίσης θέμα συγχρηματοδότηση. Το γνωρίζουμε ότι υφίσταται ως πρόταση, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο για χώρες να συνεισφέρουν από πλευράς τους σε μια περίοδο δημοσιονομικής κρίσης. Υπάρχει δυνατότητα να δράσουμε ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα, οι απασχολούμενοι να λαμβάνονται υπόψη και έτσι χρηματοδοτικά να συνεκτιμάται τι αυτό συνεπάγεται ως συνεισφορά. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να παραμείνει στο εύρος και ε, στον όγκο τον χρηματοδοτικό ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Τσουρινάν και η κυρία Κόντς. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τις ε, προκλήσεις που είπατε ότι έχουμε. Κανείς πιστεύω δεν διαφωνεί. Αναρωτιέμαι όμως ε, για τη σύνδεση σε σχέση με τις προϋποθέσεις και τη μακροοικονομία. Αυτό ε, σχετίζεται με τη δέσμη που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Εάν θέλετε ανάπτυξη και απασχόληση, δεν καταλαβαίνω ακριβώς ε, ποιο κομμάτι αυτής της δέσμης του six pack, ε, ποιο κομμάτι από αυτά θα βοηθήσει, θα ενισχύσει την απασχόληση. Εάν έχουμε μια υπερχρεωμένη χώρα και με πολύ ψηλό έλλειμμα, δεν μπορούμε να ε, συνεχίσουμε σε περικοπές και αυτή να αρχίσει να αναπτύσσεται. Δεν λειτουργεί έτσι η ανάπτυξη. Φοβάμαι ότι θα έχουμε αρνητική επίπτωση εδώ. Το βλέπουμε ήδη στο six-pack και ε, προσφέρεται, ε, παρέχεται το ίδιο, την ίδια τακτική με το six Πιστεύω ότι ίσως δεν είναι το, καλό, το σωστό φάρμακο αυτό. Πολλά ενδιαφέροντα σημεία τονίζεται για το κοινωνικό ταμείο και για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι πολύ θετικό. Η Ελίζαμπεθ είναι η εμπειρογνώμονάς μας για τα ταμεία από τους πράσινους. Ωστόσο θα πρέπει πιστεύω να έχουμε μια σωστή στρατηγική αναδιάρθρωση της Ευρώπης για να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Κίνγκα στο πολύ σύντομα κάποιες παρατηρήσεις. Η διοικητική απλούστευση και ε, μικρότερη γραφειοκρατική επιβάνηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι κάτι καλό, καλοδεχούμενο. Θα έπρεπε να ασκήσουμε πίεση όμως στα κράτη-μέλη, να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τους από πλευρά τους στον πλήρη βαθμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κανονισμοί και κανόνες ώστε τα λειτουργικά προγράμματα ουσιαστικά να ευθυγραμμίζονται και να συμμορφώνονται με τους στόχους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Και αυτή η ε, εξέλιξη δεν θα πρέπει να μας κάνει να παρακλίνουμε δηλαδή η γραφειοκρατική συρρήκνωση. Σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχθούμε σε σχέση με τις δράσεις, ε, για παράδειγμα, για τους κοινωνικά αποκλεισμένους ή τους τσιγκάνους. Θα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε κατά της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης, κατά του αποκλεισμού. Χρειάζονται ναι μεν όροι και προϋποθέσεις, αλλά όχι έτσι τελεσίδικα όπως εσύ το προτείνετε. Η περιπλοκότητα και η συνθετότητα της στρατηγικής για τους τσιγκάνου, απουσιάζει πλήρως ο συνιστόσα και στον, στην καταπολέμηση της φτώχειας πάλι μόνο πρόοδο μπορεί να επιτευχθεί αν έχουμε στοχεύσει προς μια ανάπτυξη των υποδομών, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν βλέπω να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Και όσον αφορά το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, επεκτείνοντας το φάσμα δράσεων για τους αγρότες, ποιο είναι το νόημα όσον αφορά τις επιδοτήσεις, τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διασύνδεση εδώ και για τα καινοτόμα προγράμματα καλό είναι να δούμε η μακροοικονομική προσέγγιση να συμπεριλαμβάνεται όσον αφορά την χρηματοδότηση, αλλά οι συνιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εδώ νομίζω απουσιάζουν όσον αφορά κατάρτιση, εκπαίδευση. Τι θα γίνουν για όλα αυτά στο μέλλον, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε. Οι δερμηνείς πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε στα αγγλικά. Α, θα καλύψουν και την ερώτησή μου και μετά θα πρέπει να απαντήσετε στα αγγλικά. Κύριε Επίτροπε, εγώ είμαι ανήσυχη. Ξέρω ότι το σύνολο της δέσμης εξαρτάται από ολόκληρη την Επιτροπή. Είστε μόλι ένα μέλος από τους 27 μετά από την απόφαση της 21ης ε, Ιουλίου για τη βοήθεια στην Ελλάδα είδαμε ε, για το στοιχείο της υποστήριξης πέρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αντιπαράθεση. Δεν καταλαβαίνω πώς όταν μία χώρα έχει να αντιμετωπίσει ένα ε, σχέδιο περιορισμού των δαπανών ε, και μετά στην ίδια επιτροπή δεν δίνουμε τη δυνατότητα υποστήριξης των δραστηριοτήτων με κυρώσεις. Ε, Ξεκινώντα δεύτερον όλε αυτέ τι συζητήσει, θυμάμαι ότι ο πρώην Γενικό Διευθυντή σα είχε έρθει να μου πει ότι θα πρέπει να βγάλουμε τελείω το κοινωνικό ταμείο από τον οριζόντιο κανονισμό. Ε, στο μεταξύ, εγώ βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνο στο κοινωνικό ζήτημα να μην αντιμετωπίζεται πλέον ως κοινωνικό ζήτημα. Θα γίνει δευτερεύον σε σχέση με όλους τους υπόλοιπου στόχους. Το ζήτημα της συνοχής ε, φυσικά όλες οι περιφέρειες έχουν τεράστια ευθύνη για την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής και πρέπει να κινητοποιούνται. Ωστόσο πιστεύω ότι οι συντελεστές εδώ, οι παράγοντες εδώ έχουν αντιστραφεί. Αντί να θέτουμε το κοινωνικό ζήτημα ως τμήμα της συνοχής, θεωρούμε ότι το κοινωνικό κομμάτι είναι ένα συνοδευτικό κομμάτι της συνοχής και κυρίως όταν βλέπουμε τα δημοσιονομικά ποσά για τα οποία μιλάμε έπρεπε, είχαμε πει να αυξήσουμε το μερίδιο του κοινωνικού ταμείου στον όλο προϋπολογισμό αλλά ξαφνικά του φορτώνουμε ένα σωρό πράγματα, τους γεωργούς, έχω την εντύπωση ότι ό,τι θα κερδίσουμε από τη μια πλευρά θα το χάσουμε από την άλλη. Στον οριζόντιο κανονισμό δεν μας είπατε τίποτα. Προς το παρόν ίσως να υπάρχει εκεί μέσα η ιδέα του να μην δίνουμε στα κράτη-μέλη τα χρήματα που δεν έχουν ε, ξοδέψει στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων αλλά να το χρησιμοποιήσουμε για το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Ε, αυτή είναι η πρώτη